Good morning everybody. Καλημέρα σε όλους σας. Αρχίζουμε. Δεν είμαι προσίδα βέβαια, αλλά μ' αρέσει η ακρίβεια στο χρόνο για να φύγουμε γέρος, γιατί μερικοί από εμάς θα πάμε, ξέρετε, στη Στοχόλμη. Α, τι έχουμε. Χτες το βράδυ θα είδατε όλοι την έκθεση πεπραγμένων των συντονιστών. Υποθέτω ότι διαβάσατε κιόλας. Έχει κανεί καμία αντίρρηση για αυτό που διάβασε χθε για τόσο αποφάσισαν οι συντονιστέ. Όχι. Ωραία, εγκρίνεται έτσι λοιπόν. Και προχωρούμε στην τροποποιημένη ημερήσια διάταξη. Δώσαμε την ευκαιρία στον κύριο Μπελέτη να έρθει νωρίτερα. Έμαθα ότι είχε ένα ραντεβού με τον Βασιλιά, όχι με τον Βασιλιά, με μια πριγκίπισσα μου λένε, αλλά κάτι πάρα πολύ αξιοπρεπές. Ε, ε, ε, Πονέμι, βραβεία, μια πριγκίπισσα, ε, και εκπροσωπεί ο κύριος Μπελέτ. Χαιρετισμού λοιπόν στην πριγκίψα, πάτε να πάρετε κανένα βραβείο, αλλά να μας πείτε πρώτα για την έκθεσή σας, κύριε Μπελέτ. Ευχαριστώ πολύ. Doris. Στα αγγλικά ο κύριος Μπελέτ, αλλά θα, μιλήσω ολλανδικά τη γλώσσα μου, γιατί θα είμαι όσο γίνεται πιο συνεκτικός. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα. Μάλιστα. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σε όλους σας. Δεν σας μαθαίνω τίποτα καινούριο λέγοντάς σας πόσο σημαντικό έχει γίνει πλέον το διαδίκτυο για την κοινωνία μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την κοινωνία και για την οικονομία, ε, ώστε αν υπάρξει σοβαρή διατάραξη του διαδικτύου, θα υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα και για την κοινωνία ολόκληρη και την οικονομία. Γι' αυτό αξίζει να σταθούμε λίγο στη διακυβέρνηση, το management του ίντερνετ στην Επιτροπή μας. Δηλαδή ενδεχόμενες απειλές που μπορεί να ε, καραδοκούν. Διαβάζοντας το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, Internet Governance, the next steps, διακυβέρνηση του ίντερνετ, τα επόμενα βήματα, καταλαβαίνουμε ότι η τεχνολογία και ε, υποδομή είναι απολύτως στα χέρια ιδιωτικών εταιριών. Η βασική, επαναλαμβάνω, υποδομή, οι τεχνικές προδιαγραφές, ε, η διανομή ε, διευθύνσεων IP και τα λοιπά είναι στα χέρια του ιδιωτικού τομέα. Καταρχήν αυτό δεν είναι κακό, αλλά αυτοί οι ιδιώτες ε, ασκούν δραστηριότητες που είναι κοινού ε, γενικού συμφέροντος. Μέχρι τώρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λέει ότι μέχρι στιγμής λειτουργούσε καλά η αυτορύθμιση, αυτό το self-regulating. Self-regulation. Αλλά έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι αφού ζήσαμε αυτά που ζήσαμε στο χρηματοπιστωτικό τομέα, καλό θα ήταν και στο διαδίκτυο, στα 3W, να δούμε τι ε, γίνεται στη διακυβέρνηση και να αναλάβει περισσότερο πρωταγωνιστικό και ενεργό ρόλο το δημόσιο. Δεν εννοώ εδώ ότι κάθε μέρα όλη την τεχνική υποδομή του διαδικτύου θα πρέπει να την ασκούν ε, τα κράτη. Όχι, αυτό να παραμείνει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά κάπου το κράτος θα πρέπει να έχει λόγο, να ασχολείται με τη διακυβέρνηση. Περί τίνος πρόκειται, δεν θέλω να σας πω τα τεχνικά καθόλου. Εμείς γνωμοδοτούμε, διότι γνωρίζετε ότι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι επιτροπή βιομηχανίας, αλλά εμείς ε, από την επιτροπή μας έχουμε το λόγο μας και έχουμε γνωμοδότηση να κάνουμε. Ε, θα πρέπει λοιπόν να πούμε για την παγκόσμια διακυβέρνηση του διαδικτύου ότι είναι στα χέρια του ICANN. ICAN λέγεται, Internet Cooperation for Assigned Names and, ε, και είναι αμερικανική εταιρεία με έδρα τη ε, Καλιφόρνια και υπόλογη μόνο στους νόμους της Καλιφόρνιας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το καιρό είναι στη Συμβουλευτική Επιτροπή, ε, στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο αυτής της ICAN, αλλά μέχρι εκεί είναι η συμμετοχή μας και η επιρροή μας. Το έγγραφο λοιπόν της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι ανακοίνωση εστιάζει σε αυτό το ICAN και σε αυτή τη δομή πώς ε, λειτουργεί, ε, πώς κυβερνάει το διαδίκτυο, ποια είναι η κατάσταση των πραγμάτων και τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βράχει πρόθεσμα. Υπάρχουν κάποιες βασικές προδιαγραφές βεβαίω που θέτουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει πραγματικότητα. Ε, τι εννοώ, ισόρροπη και διαφανή εποπτεία του ICAN, τι γίνεται με την ιδιωτική σφαίρα, τι γίνεται με τη διαχείριση Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι υπόλογη μόνο όχι ε, στους νόμους των ΗΠΑ, αλλά στους νόμους της πολιτείας της Καλιφόρνιας. Είναι πάρα πολύ περιορισμένη λοιπόν η δική μας επιρροή εκεί και ο έλεγχος και η υποπτία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Και εκεί είναι και η μεγαλύτερη ευαισθησία μας ε, είναι τόσο ευάλωτη ε, ακριβώς αυτή η υπόθεση, γιατί αν καταρρεύσει το διαδίκτυο θα είναι τραγικό, θα είναι πολύ κρίσιμο για την κοινωνία και για την οικονομία. Εμείς λοιπόν, ξέρετε τι θέλουμε να έχουμε ως εχέγγυα για το ε, παγκόσμιο διαδίκτυο, ένα σταθερό ίντερνετ, ε, ασφαλές, με ελευθερία του λόγου, της έκφρασης, ε, σεβασμό της ιδιωτικής σφαίρας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολυμορφία ε, πολιτισμική. Τα ξέρετε όλα αυτά. Εκεί λοιπόν θα ήθελα να τονίσω ότι είναι η σκοπιά της δικής μας Επιτροπής. Ξέρουμε ότι θέλουμε να κάνουμε πολλά στο διαδίκτυο η παιδεία ας πούμε, πολύ σημαντικό, με την ηλεκτρονική εκμάθηση και εξ αποστάσεως ε, έχουμε νέες δυνατότητες που ανοίγονται τώρα και τεράστιες με το διαδικτύο, αλλά αυτό επίσης σημαίνει ότι στη διακυβέρνηση του διαδικτύου πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα γιατί σήμερα δεν είναι ξεκάθαρα. Εδώ μιλώ για την ποιότητα της ηλεκτρονικής ε, διδασκαλίας εκμάθησης. Θα πρέπει ο καταναλωτής εντός εισαγωγικών να ξέρει αυτό η υποπτική ύλη ότι είναι αξιόπιστη, ότι ανταποκρίνεται σε προδιαγραφές και κανόνες και στη συνέχεια πρόκειται για αναγνώριση ε, των τίτλων, ε, αναγνώριση ή μεταφορά των διδακτικών μονάδων όταν κάποιος σπουδάζει online ε, να είναι σωστά στημένα τα μαθήματα και τα τμήματα. Αυτό ήταν το πρώτο για την εκπαίδευση. Ένα δεύτερο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εδώ στην Επιτροπή μας είναι η προστασία των παιδιών και των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ε, αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο. Σας παραπέμπω στο πρόγραμμα Safer Internet, ασφαλέστερο διαδίκτυο, Μόλις ξεκίνησε όμως η διαδικασία αυτή η ευαισθητοποίηση θα πρέπει να είναι μια δουλειά έτσι, μόνιμη και ε, σίγουρα σε ό,τι αφορά και τα σχολεία και τους γονείς και οι δαιμόνες και οι καλύτερες προδιαγραφές και οι καλύτεροι κανόνες ε, που προτείνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό. Επίση και ό,τι αφορά τα παιχνίδια. Είχαμε ήδη μια έκθεση σχετικά με τα παιχνίδια και τη βία των παιχνιδιών ε, των ηλεκτρονικών στο διαδίκτυο. Αυτά λοιπόν για την ενημέρωση και των γονέων. Λοιπόν, σα είπα για την εκπαίδευση, προστασία των ανηλίκων και των παιδιών και ε, σα είπα για την ε, πολυγλωσία, την πολιτιστική πολυμορφία σήμερα. ουσιαστικά ε, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη πρόσβαση για μη λατανικούς χαρακτήρες. Κινέζικα, αραβικά και ό,τι άλλο σκεφτεί κανείς, λέει ο κύριος Μπελέτ. Δηλαδή, ό,τι δεν είναι λατινικός χαρακτήρας ξεφεύγει από το διαδίκτυο ή έχει πολύ μικρή διείζηση αυτή τη στιγμή. Όταν μιλάμε όμως για την πολυγλωσία και για την πολιτιστική ε, ποικιλομορφία, μιλάμε και για γλώσσες και ε, θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιούν και εκείνοι που δεν χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες. Υπάρχει μια συμφωνία ε, μεταξύ ICAN και των αρμοδίων αρχών για τη χρήση μη λατινικών χαρακτήρων. Ε, είναι σε πάρα πολύ ευρυϊκά στάδια ακόμα αυτή η διαδικασία. Και του επόμενους μήνες και χρόνια θα πρέπει να εστιάσουμε πολύ περισσότερο σε αυτό. Σας παραπέμπω επίσης και στην πολιτιστική ε, δημιουργία του ε, διαδικτύου. Αν δεν απατώμε, κυρία Πρόεδρε, το απόγευμα ε, έχετε μια τέτοια συνάντηση για τη δημιουργική διάσταση των έργων στο ίντερνετ. Εχθές μιλήσαμε για το Google Books και την Europeana, τη βιβλιοθήκη, την ηλεκτρονική και τα προβλήματα των gatekeepers πώς θα φτάσουμε σε αυτή την ψυχιακή μορφή και πώς θα αποφύγουμε ακριβώς τον πολιτισμό να πέσουν αυτά στα χέρια ορισμένων μονοπωλίων. Και σίγουρα δεν είναι αυτά ευρωπαϊκά τα μονοπόλια και θα έχουν ε, στα χέρια τους να διαχειρίζουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και να την καθοδηγούν μέσα από μία πύλη δικτυακή. Λοιπόν, θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα. Ε, έρχομαι στις προτάσεις τώρα και τα συμπεράσματα μου. Αυτή η μονοπωλιακή κατάσταση που ζούμε σήμερα στη διακυβέρνηση του διαδικτύου και όλοι οι κίνδυνοι που ενέχονται απαιτούν επιγόντως συζήτηση. Από τις αρχές του μηνός Υπάρχει μια νέα συμφωνία μεταξύ της ICAN που σας είπα ότι είναι ιδιωτικός φορέας ε, και του Αμερικανικού κράτους για διάφορες εγγυήσει, για διαφάνεια, για ε, ανοιχτή πρόσβαση και άλλα. Υποθέτω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το γνωρίζει και θέλω να ρωτήσω εδώ τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι σε καλύτερη θέση για να εκτιμήσει και να μας πει ποιο είναι ο αντίκτυπος της νέας συμφωνίας. Είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Μόλις αυτό το μήνα ε, τέθησε η νέα συμφωνία επαναλάβα ε, μεταξύ ICAN και ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι βήμα προς τα εμπρός, δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι νομικός, διάβασα τη συμφωνία, αλλά δεν μπορώ να το εκτιμήσω. Καλύτερα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει. Και θέλω επίσης να ρωτήσω την Επιτροπή ποια είναι τα βήματα που πρέπει εμεί να κάνουμε τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να διαθέτουμε πιο ισχυρά εργαλεία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαφυλάξουμε αυτές τις αρχές που μας είναι και τόσο προσφυλείς. Συμπέρασμα τώρα, ποια είναι η ουσία. Χρειάζεται εσωτερική μεταρρύθμιση σε αυτό τον οργανισμό, τον ιδιωτικό, τον ICAN, για να υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Και ο καθένας να είναι υπόλογο εκεί, όχι μόνο απέναντι στι αρχέ της Καλιφόρνιας, αλλά ναι, υπάρχει μια πολύ πλευρή και πολυμερής ε, προσέγγιση. Πώς θα γίνει αυτό. Ε, μόνο αν ξεκινήσουμε συζήτηση με την Αμερικανική κυβέρνηση. Και με χαρά εδώ σας αναφέρω ε, αυτά που είπε η Επίτροπος κυρία Ρέντινγκ που είναι σήμερα αρμόδια για αυτά τα θέματα έχει κάνει κάποιες προτάσεις για ένα διαδίκτυο πιο διαφανές στη διακυβέρνησή του με μεγαλύτερη ευθύνη και επίση ε, δίνει μια ιδέα ενός G12. Τι είναι αυτό, ε, μια δομή ε, πολυμερής που θα επιβλέπει, θα εποπτεύει, θα ελέγχει ε, και θα είναι και υπεύθυνη για τη διακυβέρνηση και θα λογοδοτεί όχι μόνο στην Καλιφόρνια, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους εταίρους ε, απανταχού της γης. Αυτά λοιπόν, να τα πούμε και στι ΗΠΑ ότι εμεί ζητούμε συμμάχου που έχουν τα ίδια μελήματα, τέτοια συμφέροντα μαζί μα. Ε, βλέπε γνωσία, βλέπε ηλεκτρονική μάθηση, προστασία των παιδιών, όλα αυτά που σα είπα προηγουμένω. Η κυρία Ρέντινγκ κάνει και μια ρητορική ερώτηση. Αρκεί άραγε μόνο η έλευση του Προέδρου Ομπάμα να αλλάξει την κατάσταση. Ε, το πρόγραμμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στα χέρια μας όπλα. Παρά μόνο την προθυμία των Αμερικανών, εάν την έχουν και αν την εκδηλώσουν, να συζητήσουμε. Αλλιώς είμαστε εκτός νηφόνους; και πάρα πολύ ευάλωτοι. και θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι αυτό προτεραιότητα για μας στους επόμενους μήνες. Καταλαβαίνετε πόσο προβληματικό είναι αυτό. Και τώρα η ιστορία με το Google και το άλλο το δημιουργικά περιεχόμενα, τα έργα, τα copyright, πνευματικά δικαιώματα είναι μια σειρά ε, ζητημάτων που μπορούν να λυθούν μόνο παγκοσμίω. Εγώ βεβαίω είμαι στη διάθεσή σα για όλε τι παρατηρήσει, τα σχόλια, ό,τι θέλετε να μου υποβάλλετε ε, για να το βάλουμε στη γνωμοδότησή μα και να τη στείλουμε στην αρμόδια επιτροπή για την έκθεση. στην Επιτροπή Βιομηχανίας, όπως σας είπα. Αυτά. Βεβαίω είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι έχετε να προτείνετε και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Ιβο. Ο κύριος Ομπάμα τι να κάνει ο άνθρωπο. Όλοι περιμένουν με το που ήρθε ο Ομπάμα να υπάρχει αλλαγή σε όλου του τομεί. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να υπολογίζουμε στον κύριο Ομπάμα παντού και πάντα. Έχει τόσα πράγματα να διορθώσει, να τακτοποιήσει. Γι' αυτό το μικρό θέμα δεν νομίζω να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για μένα όμω είναι πολύ μεγάλο θέμα. Έχω ανισχύσει λίγο, έχω θορυβηθεί με αυτά που μα είπε. Δεν είχα καταλάβει ότι σε αυτή την ιστορία της διακυβέρνηση του διαδικτύου είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από ένα καναδικό καναδικό αμερικανικό συμβούλιο που εποπτεύει. Δεν ξέρω, να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προηγουμένως. Ο κύριος Βίλιαμ Ντί και μετά τους συναδέλφους. Παρακαλώ. Μπορείτε να μας διαφωτίσετε ίσως περισσότερο. Uh, thank you very much, Chair. Thank you. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο Μπέλετ για την πολύ ακριβή σύνοψη πολλών από τα σημεία που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν ξεκινήσω να απαντάω, θα ξεκινήσω μάλλον με την τελευταία ερώτηση, γιατί είναι η πιο επίκαιρη. Αφορά στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και ICAN, την πιο πρόσφατη συμφωνία. Η ICON δημιουργήθηκε το 1998 ε, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τη μετάβαση και τον έλεγχο σε κάποιους βασικούς ε, πόρους του ίντερνετ ε, πέραν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις ιδιωτικές εταιρείε και θέλαμε να υπάρχει διεθνής εκπροσώπηση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στήριξε ολόψυχα Τότε ήταν η κυβέρνηση Κλίντον και έκανε αυτή την απόπειρα να επιτύχει αυτόν τον στόχο. Το διαδίκτυο φυσικά είναι προς το ενδιαφέρον όλων των πολιτών και θα ήταν ε, ε αδύνατον μία κυβέρνηση να ασκεί εποπτεία σε ένα, ε, στο διαδίκτυο το οποίο μας αφορά όλους παγκοσμίως. Τα κράτη-μέλη συμμετέχουν στην Επιτροπή Κυβερνήσεων, η οποία είναι μια επιτροπή που δίνει συμβουλές προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ICAN και θέλουν να δούνε τι γίνεται με τους στόχους δημόσιας Πολιτική για το διαδίκτυο. Από το 1998, ε, στα πλαίσια της μετάβασης, έγιναν διάφορες διμερείς συμφωνίε μεταξύ τη κυβέρνηση των ΗΠΑ και τη ICAN και πρέπει να πω ότι υπάρχει ένας κάποιος βαθμός απογοήτευσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι αυτές οι διμερείς συμφωνίες εξακολουθούν να ισχύουν πολύ καιρό μετά. Αρχικώ είχαμε θεωρήσει ότι αυτέ οι διμερεί συμφωνίε είναι μεταβατικό μέτρο, αλλά μετά από τόσα χρόνια εξακολουθούν να ισχύουν. Η νέα συμφωνία θεωρούμε ότι είναι θετικό στοιχείο, ένα θετικό δείγμα, διότι αυτή η κυβέρνηση η οποία υπάρχει πλέον στην Ουάσιγκτον ε, φαίνεται να στρέφεται προς την Ευρώπη. Κάλεσαν το Ιντρόικα των Προεδριών για επίσκεψη στην Ουάσιγκτον το Σεπτέμβριο για να ακούσουν και τις απόψεις μας για το πώς νομίζουμε ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί μελλοντικά η ICAN και πώς θα πρέπει ε, να ληφθεί υπόψη και η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρούμε ότι στην τελευταία συνεδρίαση ελήφθησαν υπόψη πολλά από τα στοιχεία που τους είπαμε. Υπάρχει πιο συγκεκριμένη μνήμα στην ανάγκη ε, η ICAN να είναι παγκοσμίου ενδιαφέροντος και επίσης αναγνωρίζεται και το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να διαδραματίσουν πολύ συγκεκριμένο ρόλο στην διαφύλαξη των δημοσίων συμφερόντων σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι το σημείο αυτό είναι σημαντικό. Μέχρι τούδε όλοι ε, ευρύτατα αναγνώριζαν ότι το διαδίκτυο αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς καμία άμεση ε, συμμετοχή κυβερνήσεων. Και αυτό δεν είναι σύμπτωση. Υπήρξαν πάρα πολλές πρωτοβουλίε από ακαδημαϊκούς κύκλους, από ιδιωτικούς κύκλους και όλοι υποφοληθήκαμε από αυτή τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1,5 ε, δις χρήστες του διαδικτύου. Πολύ ε, σύντομα θα αυξηθούν ακόμα πολύ περισσότερο, κυρίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και η αθρώα πλειονότητα των χρηστών του διαδικτύου δεν συμμετέχουν σε κανέναν ε, από τους φορείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή αποφασίζουν για το διαδίκτυο. Οι περισσότεροι από τους χρήστες δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή τους. Έτσι είναι τα πράγματα, απλά. Επομένως, Οι χρήστε του διαδικτύου, είτε πρόκειται για ε, ατομικού χρήστε ή επιχειρήσει, ε, ε, περιμένουν λογικά οι κυβερνήσει να προασπίζουν τα συμφέροντά του. Ένα φορέα λοιπόν σαν τον ICAN είναι ένα ε, πολυμερή φορέα, έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή από ιδιωτικού φορεί, έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή από την κοινωνία των πολιτών και έχει και έναν εκπληκτικά μεγάλο αριθμό κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη GAC την Επιτροπή των Κυβερνήσεων. Αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο δραστηριοί για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τη δημόσια πολιτική και να μην ανταποκρινόμαστε απλά στα προβλήματα όταν προκύπτουν. Και αυτό είναι το βασικό θέμα της ανακοίνωσης, το οποίο πολύ σωστά ε, αναφέρατε. Τώρα, για να επανέλθω στη συμφωνία, να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι αυτή είναι μια διμερή συμφωνία μεταξύ ΙΠΑ και ΆΙΚΑΝ. Αυτοί είναι οι δύο συνυπογράφοντε. Καμία άλλη κυβέρνηση, εξ όσων γνωρίζουμε εμεί, δεν συμμετείχε στην ε, ε, προετοιμασία αυτής της ε, συμφωνίας. Δυστυχώ προς το παρόν αφορά εσωτερικά θέματα των ΙΠΑ Ε, υπάρχει βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλά από τα πράγματα που αναφέρονται είναι πολύ καθησυχαστικά, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι μέλη γενέστε και πώς θα εφαρμοστεί. Στόχος είναι να δημιουργηθούν και ε, πάνελ αναθεώρησης για να εξετάσουν την απόδοση του ΣΑΙΚΑΝ ως προς τα θέματα διαφάνειας, ε, του σε ποιον είναι υπόλογοι, αν είναι υπόλογοι στη διεθνή κοινότητα. Και το πρώτο πάνελ Ελπίζουμε να ξεκινήσει στις αρχές ε, του νέου έτους και να έχουμε και την πρώτη έκθεση μέχρι το τέλος του 2010. Εμείς ερμηνεύουμε αυτή τη συμφωνία ε, και νομίζω ότι αυτή την άποψη συμφωνούν και είπα, ε, ω προ το ότι θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή από πλευρό κυβερνήσεων για τι δραστηριότητε και, και την εποπτεία τη ICAN. η αναθεώρηση της ICAN γίνεται ουσιαστικά από τους ανθρώπους της ICAN, από όλους αυτούς που έχουν μεγάλα εμπορικά συμφέροντα στη διαδικασία και αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνη για τα βασικά στοιχεία της ε, διαδικασίας πολιτικής της ICAN. Εμείς αυτή τη στιγμή πιέζουμε, πιέζουμε πάρα πολύ προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη συμμετοχή της κυβέρνησης ε, στα πάνελ όπως λέτε πολύ σωστά, δεν ε, φροντίζουμε πάρα πολύ το διαδίκτυο και τα πάνελ αναθεώρησης, αλλά αν είναι να νομιμοποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κυβερνήσεις να εκπροσωπούνται στι επιτροπές αυτές. Δεν μπορούμε να έχουμε μία μονομερή κατάσταση και να έχουμε ε, πάνω από 200 κυβερνήσεις σε κάθε μία από τις ε, επιτροπές αναθεώρησης, θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη γεωγραφική εκπροσώπηση και πολιτική εκπροσώπηση, ώστε να προσδώσουμε νομιμότητα σε όλη αυτή τη διαδικασία αναθεώρησης και από πλευράς δημόσιας πολιτικής να υπάρχει και ε, η ασφάλεια ότι όντως στηρούνται αυτοί οι στόχοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσω εδώ. Δεν ξέρω αν θέλουν κάποιοι άλλοι ε, συνάδελφοι ευρωβουλευτέ να μιλήσουν. Ε, με χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ομολογώ ότι μπερδεύτηκα ακόμα περισσότερο από ότι ήμουν προηγουμένω. Λοιπόν, τι να σας πω. Δεν ξέρω τι να πταίει. Αλλά μου φαίνονται όλα αυτά πάρα πολύ αδιαφανή και πάρα πολύ μυστήρια και πάρα πολύ περίεργα. Και πώς είναι δυνατόν να υπάρχει συμφωνία μεταξύ ΆΙΚΑΝ και Αμερικής και να κάνουν μεταξύ τους συμφωνίες και πλακάκια για ένα θέμα που μας αφορά όλους μας. Πραγματικά αυτό αδυνατό να το καταλάβω. Και τι είναι αυτή η Επιτροπή Διακυβέρνησης. Ποιο να συμβουλεύει, ποιε κυβερνήσεις. Λεφτά τίποτα συμμετέχουμε Εμεί οικονομικά. Μπορείτε να μας πείτε δύο προτάσεις να μας εξηγήσετε. Δεν έχω καταλάβει. Yes, and I apologize for not being clearer before. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν αρκετά σαφής. This is actually a very um, uh, complex area with a very unusual history. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα και είναι πολύ περίεργη και η εξέλιξή της. Μιλάμε για την εκχώρηση αριθμών και διευθύνσεων. Είναι τα domain names που γνωρίζετε όλοι, για παράδειγμα ε, europa.eu, καθώς επίσης και τις ε, διευθύνσεις που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές για να έχονται σε επαφή ο ένας με τον άλλον. Αυτό το σύστημα αναπτύχθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες από πανεπιστημιακούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 αποφασίστηκε ότι... Ε, δεν θα έπρεπε αυτοί οι πόροι να διαχειρίζονται από ακαδημαϊκούς ε, σε part-time μάλιστα. Αποφασίστηκαν λοιπόν οι πανεπιστημιακοί και οι κυβερνήσει που συμμετείχαν, γιατί όλα αυτά ήταν τμήμα χρηματοδότηση, όλα αυτά μεταβατικά να περάσουν σε ε, μια οργάνωση του ιδιωτικού τομέα. Στη διαδικασία όμως της ιδιωτικοποίησης, οι Ηνωμένε Πολιτείε έκαναν ένα μνημόνιο συνεννόησης με την ICAN και υπέγραψε και μια σχετική σύμβαση για τη διαχείριση των πόρων και για ιστορικούς λόγους έχουμε λοιπόν την έδρα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Από εκεί και πέρα η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να διεθνοποιήσει εντός εισαγωγικών αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει μόνιμη δέσμευση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να το εξετάσει και να κάνει κάτι με το θέμα, αλλά με την, τελευταία, με την προηγούμενη κυβέρνηση υπήρξε πάρα πολύ μικρή πρόοδος Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή μια ιστορική ευκαιρία στα χέρια μας με τη νέα κυβέρνηση να τους προσπαθήσουμε να τους πιέσουμε να τηρήσουν τη δέσμευση που είχε αναλάβει η προηγούμενη δημοκρατική κυβέρνηση και να μπει στο θέμα στη διεθνή αρένα. Αλλά θα είναι δύσκολο. Όσον αφορά στη δική μας συμμετοχή, εμείς συμμετέχουμε ε, χωρίς χρηματοδότηση. Πληρώνουμε τη συμμετοχή μας σε αυτές τις δραστηριότητες Γίνονται τρεις συνεδριάσεις ετησίων, τρεις δημόσιες συνεδριάσεις, ε, συνήθως σε διάφορα μέρη ανά τον κόσμο. Επομένως είναι και ακριβά, αρκετά δαπανηρή η διαδικασία για να συμμετέχουν οι κυβερνήσεις, αλλά δεν συνεισφέρουμε χρηματοδοτικά, χρηματοδοτούνται από τον ιδιωτικό τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ποιο θέλει από τους συναδέλφους να μιλήσει για αυτό το τόσο περίπλοκο θέμα. Παρακαλώ, κύριος Βάτιμο. Συγγνώμη. Εγώ καθυστέρησα λίγο να έρθω, αλλά αρχίζω να μην γνωρίζω τι είναι η ICAN. Τι σημαίνει η ICAN. Αυτό το πράγμα το οποίο συζητάτε συνεχώς. Ναι, στην αρχή το είπαμε κύριε Βάτιμο, να σας διαβάσω τι λέει εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στο ΚΑΚ, στο ICAN. Τι είναι το ICAN τώρα. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Δίνει διευθύνσεις και ονόματα και αριθμούς. Αυτό είναι. Μάλιστα. Anybody interested? Άλλος κανείς που να ενδιαφέρεται να πάρει το λόγο. Ποιος? Α, ο κύριος Μπίσκι, παρακαλώ. Μια ερώτηση έχω. Τι, ποιες αρακτικές θα είχαμε δηλαδή με το ιδιωτικό καθεστώς και το δίκαιο της Καλιφόρνιας δεν πήγαν και τόσο άσχημα τα πράγματα. Ποιες θα ήταν οι εναλλακτικέ λύσεις έτσι ώστε να συμμετέχουν, ξέρω εγώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών. Γιατί στο Δίνεκες δεν επιτρέπεται τέτοια κατάσταση να περνάνε όλα από τα χέρια ιδιωτικών εταιριών. Είναι δημόσιο αγαθό. Μπορεί κανείς να το οργανώνει ε, ιδιωτικά και δεν χρειάζεται να δαιμονοποιούμε την ΙΚΑΝ. Έχει και πολλά καλά. Αλλά ποιε είναι οι εναλλακτικέ λύσει και τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω και εγώ ερώτηση, λέει η κυρία Πακ. Αν δεν θέλει κανένα συνάδελφο να ρωτήσει τίποτα άλλο. Ο Ήβο επέμεινε πάρα πολύ στο θέμα άλλου χαρακτήρε, πλην λατινικών. Μα και στην Ευρώπη έχουμε κυριλικά. Ε, υπάρχουν τα κυριλικά ε, εκεί πέρα όπως και τα λατινικά. Τι μόνο τα κινέζικα είναι τα ιαπωνέζικα που έχουν πρόβλημα η κυριλικά και άλλες γραφές, λέει η πρόεδρος. Αυτά είχα να ρωτήσω κι εγώ. Η κυρία Ράμπ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ έχω μια ερώτηση και πάλι για τις εναλλακτικέ προτάσεις. Μιλήσατε, κύριε Μπελέτ, για την κυρία Ρέντινγκ που προτείνει μια δομή του G12, δηλαδή με πολλά μέρη και πολλού πόλου, Ποιοι θα ήταν αυτοί λοιπόν που θα συμμετείχαν εκεί στην G12. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόρις. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση για το e-learning. Εξ εκπαίδευση. Προβλέπονται κάποια κονδύλια για να υποστηρίξουμε το σχετικό σύστημα. Με ταυτόχρονη διασφάλιση ποιότητας. Επομένως, ε, θα πρέπει με τα κονδύλια αυτά να προάγονται και τα συστήματα. Πολλά κράτη-μέλη έχουν ε, πρόσβαση. Κατά την άποψή σας υπάρχουν δυνατότητες να υποστηριχθεί αυτή η πλατφόρμα του e-learning. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ. Ε, μια πρόταση μόνο. Πολλοί έχουμε προβλήματα με την ICAN από μας και ανασφάλειες. Δεν θα μπορούσαμε για επόμενη συνεδρίαση να καλέσουμε εξωτερικό εμπειρογνώμο να μας μιλήσει μισή ώρα για το υπόβαθρο και τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί και με τα νέα μέσα θα το βρούμε μπροστά μας. Η Πρόεδρος. Εμεί πάντα στέλνουμε κυρίους και κυρίες ε, σε αυτά τα όργανα. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπάρχει κανείς που να ασχολήθηκε εντατικά με αυτό το θέμα να έρθει να μας ενημερώσει. Να μας κάνει μια μικρή διάλυση. Λίγο περισσότερα από αυτά που μας είπατε σήμερα εσείς ε, από την Επιτροπή. Έτσι. Η κυρία Χάνιμπαλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσο προχωράμε σε αυτό το θέμα τόσο πιο περίπλοκα γίνονται τα πράγματα μου φαίνεται. Και φαίνεται να είναι κάτι το οποίο πάει πολύ πίσω. Και εμεί ουσιαστικά δεν είχαμε καμία συμμετοχή και δεν φαίνεται να έχουμε και καμία δυνατότητα να συμμετάσχουμε. Διορθώστε με αν κάνω λάθο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι λίγο θολά τα πράγματα. Θα ήθελα και κάποιε επιπλέον πληροφορίε, είμαι υπέρ αυτού και ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε και πώς μπορούμε να το προσεγγίσουμε από ευρωπαϊκής προπτικής και να πάρουμε αυτά τα οποία συζητάμε, να περάσουμε τα μηνύματά μας, να υπάρχει μια στρατηγική προκειμένου να καταλήξουμε για κάπου με όλο αυτό το πράγμα. Διότι μου φαίνεται ότι θα είναι τεράστια η δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένας κάποιος στόχος στο τέλος, μια ηθάκη. Σε ε, thank you very much. similarly. Ευχαριστώ. Μήπως θα μπορούσε να μας συνοψίσει σε μια-δυο προτάσεις ε, ποιος είναι ο τελικός μας στόχος, τι προσπαθούμε να επιτύχουμε με όλα αυτά, αν δεν είναι τόσο περίπλοκο. Ευχαριστώ πολύ. das wird ein bisschen schwierig Α, εδώ λίγο δύσκολο το πράγμα, διότι εμείς γνωμοδοτούμε και μόνο. Επί της ουσίας αρμόδια είναι Επιτροπή Βιομηχανίας. Αν απαντήσει ο Ήβος στις ερωτήσεις θα δούμε και πολύ σύντομα και σε αυτό που ρώτησε ο κύριο Κέλλη. Ορίστε, Ιβο Μπελέτ. Ναι. Σα ευχαριστώ πολύ. Να τα πω δικά. Είναι πιο εύκολο για μένα, γιατί είναι περίπλοκα τα πράγματα. Και να ακούσουμε ξανά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν χρειάζεται, γιατί και εγώ τεχνικός δεν είμαι σε αυτά τα θέματα και ειδικό. Τις τελευταίες εβδομάδες διάβασα πάρα πολλά για αυτά τα θέματα, αλλά παραμένουν πολύ τεχνικά. Πρώτα απ' όλα να σα απαντήσω στο εξή. Βεβαίω δεν υπάρχει άμεσο κίνδυνο αυτό που λέει ο κύριο Μπίσκι. Εντάξει, ναι. Λειτουργεί το διαδίκτυο, έχει τόσο μεγάλη επιτυχία ε, και έχει και ε, πολύ καλή διακυβέρνηση. Και αυτό επιτυχία είναι. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα πάνε ρολόι. Το είπα από την αρχή. Στόχο δεν είναι να το πάρουμε από τον ιδιώτη για να το έχουμε εμεί στα χέρια μα, να το δώσουμε στο κράτο. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε τέτοια πρόθεση εμεί για να μην πω ότι δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ό,τι κατάλαβα έχει τέτοιε προθέσει. Αλλά επειδή δεν υπάρχει σήμερα πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι στο επόμενο ε, διάστημα, στο άμεσο, προσεχέ μέλλον, δεν θα προκύψει κανένα πρόβλημα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητα όλα αυτά τα πράγματα. Αν διαβάσετε την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM 2009, ε, ε, εννιά σελίδε είναι, δεν είναι μεγάλο. Καταλάβετε τι είναι AI. Δεν χρειάζεται να είσαι τεχνικό για να το καταλάβει. Και θα δείτε και πόσο εύθραυστα είναι τα πάντα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί εστιάζει. Βέβαια, με την Επιτροπή Βιομηχανία, αν διαβάσετε το έγγραφο, θα καταλάβετε την ανακοίνωση Επιτροπή. Αλλά είναι πολύ σημαντικέ οι αρχέ και ε, οι φάκελοι και τα ζητήματα σας είπα. Google Books, προστασία των παιδιών, πολυγνωσία. Ε, ε, όλα αυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα. Δεν τα γράφει αυτά ο φάκελο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ σα τα ανέφερα ω παραδείγματα γιατί δικό μα ρόλο τη δική μα Επιτροπή Πολιτισμού, Εκπαίδευση, Νεολαία είναι αυτό που μα ενδιαφέρει. Άλλο το κεφάλαιο τη βιομηχανία και τη ουσία. Έτσι, δεν παραπέμπω άμεσα στο έγγραφο. Τι είναι το endgame που λέει ο Σον Κέλλη, Ποιο είναι ο στόχο και τι επιδιώκουμε. Επανέρχομαι στην πρόταση της κυρίας Ρέντινγκ πριν από μερικού μήνε. Ε, είπαμε ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να έχουμε περισσότερο λέγινε και περισσότερη επιρροή, να συμμετέχουμε. Γιατί τώρα είμαστε σε αυτό το συμβουλευτικό όργανο, αλλά τι πράγμα, αυτό τίποτα. Εντάξει, δίνει συμβουλές θα πρέπει να περάσουμε σε μια πολυμερή διαχείριση του ε, παγκοσμίου ιστού. Ε, γι' αυτό προτείνει η, πρόεδρος, με, η, κυρία Ρέντινγκ συγγνώμη, με το G12. Ποιοι να συμμετέχουν εκεί, οι μεγάλοι εταίροι παγκοσμίω. Οι Αμερικανοί που έτσι και αλλιώ είναι εκεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω εγώ, Κίνα, Ινδία. Μια σταδιακή εκπροσώπηση εκεί Κάνουν προτάσει εκεί ενδεχομένω. Ενδεχομένω. Από πού να τι κάνουμε, από τον ΟΗΕ. Στον ΟΗΕ μόνο αυτό του έλειπε. Είναι τεράστιο μηχανισμό, ε, τεράστια δομή. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να έχουμε μία δομή ακριβώς επί τούτου, αυτό το G12 ας πούμε, που να διαπραγματεύεται άμεσα για την ε, ηλεκτρονική εκμάθηση, το e-learning και Νομίζω ότι υπάρχουν ήδη προγράμματα γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας διαφωτίσει περισσότερο για το e-learning και την υποστήριξή του. Υπάρχει μεν, αλλά αυτό δεν αφαιρεί καθόλου ε, το γεγονό των απειλών. Δηλαδή, ε, πραγματικά καραδοκούν και πάλι εταιρείε ή ξέρω, πανεπιστήμια για τη διαφύλαξη της ποιότητας, για τους τίτλους που απονέμονται και τα πτυχία, ε, τις ισοτιμίες και αυτό που λέτε πρόεδρε και εσείς για την πολυγλωσία και τους μη λατινικούς χαρακτήρες, ε, αν κατάλαβα καλά, μπορεί να με διορθώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ασφάλω, αρχές Νοεμβρίου προβλέπετε ότι μπορεί να ανοίξει ICAN και για άλλους χαρακτήρες, για άλλα αλφάβητα που δεν είναι λατινικά. Κυρικά, αραβικά και κινέζικα. Εξ όσων γνωρίζουν, πρόκειται για όλους τους μη λατινικούς χαρακτήρες. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μια συμφωνία στα χαρτιά εφαρμόζεται την άλλη μέρα. Μπορεί να χρειαστεί πάρα πολύ καιρό. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην Αφρική και στην Ασία. Αυτά. Έτσι, ε, με λίγα λόγια, υποθέτω ότι μπορεί να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Κύριε Ντί, θα μπορούσα να σας ξαναδώσω το λόγο για να απαντήσει σε ερωτήσεις. Και αυτό που προτείνει η κυρία Ρέντινγκ και θα αναλάβει μάλλον τώρα η κυρία Κρός, τι σημαίνει, μπορούμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε συμφωνία με την ICAN, όπως έχουν και οι Αμερικανοί ή κάτι τέτοιο. Παρακαλώ. Um, thank you. Um... Ευχαριστώ. Δεν θα μπορούσα ποτέ να διανοηθώ να μιλήσω εξ ονόματος του Επιτρόπου μου. Όταν έγιναν αυτά τα σχόλια από πλευρά τη κυρία Ρέντινγκ, ήταν μια απόπειρα να προσπαθήσουν να προλάβουν κάποια συζήτηση επί του θέματο. Υπήρχε και ένα άγχο από πλευρά τη ότι θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε νέα συμφωνία χωρί δημόσια συζήτηση επί του θέματο. Και νομίζω ότι ήταν επιτυχέ αυτό. Και φαίνεται και αυτό και από την αντίδραση που είχαμε. Κατά την άποψή μου, η νέα συμφωνία μεταξύ ICAN και ΙΠΑ ε, συμπεριλαμβάνει κάποια στοιχεία του G12. Θα πρέπει βέβαια να δούμε ε, πώς μπορεί να τα εφαρμόσει αυτά στα πάνελ αναθεώρησης. Αν τα εφαρμόσουν με τρόπο ώστε να υπάρχει μεγάλη εκπροσώπηση από γεωγραφικής πλευράς ε, για τους χρήστες του διαδικτύου, ίσως να μπορέσουμε να το θεωρήσουμε ένα μεταβατικό βήμα ως προς την πορεία για μια πιο καλή λύση. Προς το παρόν όμως η ICAN εξακολουθεί να είναι εντός των ιδιωτικών οργανώσεων. Στην ε, διάρκεια μεταξύ του 2000, της ε, Παγκόσμιας Διάσκεψης για το 2003 έως 2005 ε, το θέμα ήταν ένα από τα φλέγοντα ζητήματα, εξετάστηκε επισταμένος, υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις επ' αυτού, αλλά υπήρχε μια μεγάλη διάσταση απόψεων μεταξύ εκείνων που θέλουν να συνεχίσει να λειτουργεί το διαδίκτυο χωρίς κυβερνητική παρέμβαση και εκείνων που πιστεύουν ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των κυβερνήσεων ώστε να διασφαλίσουμε ότι επιτυγχάνονται και οι στόχοι δημόσιας πολιτικής. Τα Ηνωμένα Έθνη και η ITU, η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, είπαν ότι θα μπορούσαν ίσως αυτοί να αναλάβουν τις ε, αρμοδιότητες της ICAN και αυτό προκάλεσε μια πάρα πολύ στεναρή αρνητική αντίδραση από πολλές ε, δυτικές ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και αρκετών ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιστάθηκαν στεναρά και αυτό φυσικά μας οδήγησε και στο ερώτημα το οποίο είναι ακόμα σε κρεμότητα. Πώς μπορούμε να έχουμε μία πολυμερή συμφωνία που θα περιλαμβάνει τους πάντες και θα σέβεται τα δικαιώματα κάθε χώρα ανά τον κόσμο για να ε, εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του διαδικτύου χωρίς να υπάρχει ε, και ένας δημόσιος φορέας. Εξακολουθεί να εκκρεμεί λοιπόν αυτό το ερώτημα και δεν νομίζω ότι η λύση είναι να πούμε ότι εμείς δεν έχουμε λύση, επομένως απομακρυνόμαστε από αυτό το πρόβλημα. Ε, πολλοί λένε ότι αν δεν μπορείτε να πείτε ακριβώς τι μοντέλο θέλετε να προτείνετε, δεν θα πρέπει καν να θέτετε το πρόβλημα. Ε, νομίζω ότι είναι μια πολυμερή διαδικασία. Ε, πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνομιλούμε με τους διεθνείς εταίρους μας προκειμένου να εξεύρουμε κάποια λύση και να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις ώστε το θέμα να μην εξαφανιστεί και να θεωρούν ότι όλοι, όλα είναι καλά, υπάρχει μια κυβέρνηση που ασκεί μονομερή έλεγχο και όλα εντάξει. Το θέμα λοιπόν είναι πολύ προφανές, η απάντησή του δεν είναι τόσο προφανής. Νομίζω ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μέχρι τούδε είναι ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να το συζητούμε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να συζητούμε με τους διεθνείς εταίρους μας και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και ευρωπαϊκή συνένεση επί του θέματος. Διότι ε, στο παρελθόν όταν κάναμε διεθνείς συζητήσεις δεν ήταν πάντα σαφές ότι υπάρχει σαφή, ε, συνένεση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος. Και αυτό φυσικά ε, μας δημιουργεί και ε, μια μειονεκτική θέση, αν θέλετε, διότι δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε ως μια φωνή. Τώρα, για το να γίνουν διεθνή τα domain names, ε, να μπορεί κάποιος δηλαδή να εγγράψει ένα όνομα χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο τρόπο γραφής που δεν είναι λατινικός, για παράδειγμα. Όταν γράφετε κάτι, το ε, europa.eu, το EU είναι domain υψηλού επίπεδου και αυτό μπορούν να το διαχειριστούν. Το υπόλοιπο προσφέρει τη δυνατότητα ε, εδώ και ένα-δύο χρόνια να χρησιμοποιούνται και άλλοι χαρακτήρες. Αυτό λοιπόν έχει ήδη εισαχθεί διεθνώς. Γιατί ήταν πολύ σημαντική η ανακοίνωση της ICARS και γιατί την χαιρετίζουμε, είναι γιατί άρχισαν να δέχονται αιτήσει από χώρε που θέλουν να συμπεριλάβουν και το τελευταίο κομμάτι, παραδείγματο χάρη, το τελεία CN αυτή τη στιγμή είναι για την Κίνα, αλλά το CN είναι ένα λατινικό συνδυασμό χαρακτήρων. Επομένω, οι Κινέζοι θα πρέπει να μπορούν να βάλουν ε, ένα domain ε, top level στον βασικό του χαρακτήρα στα κινέζικα, ώστε να είναι όλο το όνομα σε κινέζικο αλφάβητο, να έχετε και αραβικά, ε, ινδικά. Ότι... Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους χρήστες του διαδικτύου που δεν χρησιμοποιούν λατινικό αλφάβητο στη γλώσσα τους. Μα χαροποιεί λοιπόν ιδιαίτερα και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη στο διαδίκτυο και ικανοποιεί τους πάντες. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Ε, Ευχαριστώ. Η συζήτηση αυτή ήταν σημαντική και διαφωτιστική μέρη και μέρη μας οδήγησε σε μεγαλύτερη σύγχυση. Νομίζω θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα με τον Ήβο και μάλιστα εντατικά το ξανασυζητήσουμε. Να κοιτάξουμε τι γίνεται και στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Γιατί είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε και τις απόψεις και την προσέγγιση της βιομηχανίας, αν εντοπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμά, ας πούμε. Έτσι, από τη σκοπιά του πολιτισμού, που εμείς δεν είμαστε η τεχνική της υπόθεσης και η ειδική. Ωραία. Δεν κλείνει εδώ το θέμα, έχουμε πολλά ακόμα. 26 Ιανουαρίου ο κύριος Μπελέτ θα μας φέρει το σχέδιο γνωμοδότησή του και στις 22 Φλεβάρι πλέον 22 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ήβο. Καλή διασκέδαση με την πριγκίπισσα. Και πάμε στο επόμενο θέμα στη Μέση διάταξη. Er Στην πριγκίπισσα, το είπα και προηγουμένως. Τι να σας πω. Δεν ήσασταν όλοι παρόντες. Λοιπόν, πάμε στο 7. Τι λέει εδώ. Έχουμε εδώ τον κύριο Ρίτσαρτ Ντόχερτη που θα μας παρουσιάσει μια μελέτη με θέμα η μελλοντική κατεύθυνση της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία. Θα χρησιμοποιήσει μάλιστα και το διαδίκτυο για το σκοπό αυτό. Παρακαλώ, κύριε Ντόχερτη. Συγγνώμη. Καλημέρα σε όλους. Έχω ετοιμάσει εδώ μια μικρή παρουσίαση, η οποία σας διανέμεται τώρα και θα μπορείτε να τα δείτε και στις οθόνες σας νομίζω. Αυτή η σύντομη εισαγωγή λοιπόν από πλευρά μου είναι απάντηση σε ένα αίτημα το οποίο λάβαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας κάνουμε μια μικρή αναλυτική μελέτη για την κατάσταση της ε, πολιτικής για τη νεολαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ επίκαιρη αυτή η παρουσίαση. Πρώτον, για την περασμένη Παρασκευή το Συμβούλιο υιοθέτησε το τελευταίο του, την τελευταία του ανακοίνωση για το θέμα αυτό, σε μια σειρά από πολύ σημαντικά βήματα τα οποία γίνονται επί του θέματος. Και δεύτερον, θα γνωρίζετε όλοι ότι από σήμερα και στο εξή ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνα. Και αυτό ε, σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές ε, συνέπειες για το θέμα αυτό. Θα αναφερθώ και στις δύο αυτές ε, διαστάσεις στη σύντομη παρουσίαση που θα σας κάνω. Να σας δώσω λίγο το, το υπόβαθρο και από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε τους τρεις βασικούς πυλώνες της πολιτικής για την νεολαία. Οι πυλώνες αυτοί είναι ο εξορθολογισμός και η προσέγγιση ανατομέα σε όλα τα θέματα που αφορούν στους νέους, ε, που φυσικά τους αφορούν πάρα, πολλούς, πάρα πολλοί τομείς πολιτικής. Το δεύτερο είναι η ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, ο μηχανισμός δηλαδή μέσω του οποίου ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασχοληθεί με την πολιτική και την νεολαία, διότι δεν υπάρχει επίσημη αρμοδιότητα στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διαχειρίζεται την πολιτική. Και ο τρίτος βασικός πυλώνας είναι ο δομημένος διάλογος. Ένας διάλογος μέσω του οποίου ε, θα μπορούν να συμμετέχουν οι δημόσιες αρχές, αλλά και οι νέοι και οι ίδιες οι Με δομημένο τρόπο για την ανάπτυξη και τη συζήτηση της πολιτικής. Και επίσης θα, θα ασχοληθούμε στην τομέα με τον τομέα της έρευνας, ο οποίος ε, φυσικά διέπει την όλη ανάπτυξη πολιτικής στον τομέα αυτά και θα δούμε και λίγα πράγματα για το τι φέρνει η συνθήκη της Λισαβόνα ε, και τι νέες προοπτικές έχουμε. Να σας δώσω λίγο το ιστορικό ανέφερα την απόφαση του Συμβουλίου της περασμένης Παρασκευής. Ε, αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν εξελίξει εδώ και αρκετά χρόνια. Πριν από 20 χρόνια έγινε το πρώτο βασικό βήμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε και το Συμβούλιο υιοθέτησε το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα για τους νέους. Τότε το αποκαλούσαμε Youth for Europe. Έκτοτε είχαμε ε, μια σειρά από πιο πολιτικά βήματα, το, η κορύφωση των οποίων ήταν ε, η πολιτική για τα επόμενα εννέα χρόνια. Αναφέρθηκα στους τρεις πυλώνες, την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Νέων, το οποίο εθετήθηκε πριν από κάποια χρόνια και προχώρησε τα αρχικά βήματα και οδήγησε την ευρωπαϊκή πολιτική πιο κοντά στην ε, οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως τότε συνδέοντας τους στόχους της πολιτικής για τους νέους ε, στους βασικούς στόχους της ε, στρατηγικής της Λισαβόνας. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Νέων το υλοποίησε αυτό στα μέσα της ε, δεκαετίας μας και προσπάθησε να εξορθολογήσει τις ανησυχίες ε, για την νεολαία σε άλλες ε, πολιτικές, κυρίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε επίπεδο Γενικών Διευθυντών και με τα Υπουργεία σε εθνικό επίπεδο. In a major, um, element of the community's τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την υποστήριξη της νεολαίας ήταν πολύ βασικά και εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και το τελευταίο σημείο της ε, διαφάνειας, τη συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, δραστηριοποιείται σε θέματα νεολαίας πολύ περισσότερο καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αναπτύξει μια σειρά από προγράμματα από το τέλος του πολέμου και μετά, σε στενή συνεργασία με οργανώσεις νεολαίας, ε, με πολλές από τις χώρες που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά πριν από 20 χρόνια που άρχισε να ασχολείται με το θέμα μπόρεσε να προσφέρει πολύ περισσότερους οικονομικούς πόρους και αναπτύχθηκαν πάρα πολλά προγράμματα για τους νέους ε, στο πλαίσιο αυτό και έχουμε πλέον το πρόσφατο πρόγραμμα Youth in Actions που έχει ένα ε, προπολογισμό άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 7 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αυτή τη στιγμή δαπανά πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ε, για τις δραστηριότητες αυτές και συνεργάζεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, έχουμε συνεργασία η οποία αφορά κυρίως σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων και ε, επιμόρφωση νέων για να υποστηρίζουν τα θέματα της νεολαίας. Όσον αφορά τώρα στο νομοθετικό πλαίσιο, Αναφέρθηκα στο, στην απόφαση Συμβουλίου που υιοθετήθηκε την Παρασκευή. Αυτή είναι συνέχεια τη ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είχαμε στι αρχέ του έτου, που, ε, που συμπεριλάμβανε συγγνώμη, όλα όσα έχουμε μέχρι σήμερα για του νέου. Ε, είχαμε μια πολύ χρήσιμη έκθεση, την οποία εκπώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώ έχει κατάσταση για του νέου ε, σήμερα. Και την πρόοδο ε, την οποία επιτύχαμε με τη μέθοδο ανοιχτού συντονισμού για την εφαρμογή του Συμφώνου για την Νεολαία μέχρι σήμερα. Η νέα απόφαση ε, αποδέχεται και υλοποιεί μια νέα στρατηγική για τα επόμενα 8 χρόνια, η οποία θα υλοποιηθεί σε τρεις κύκλους των ε, τριών ετών οι προεδρίες του Συμβουλίου θα έχουν μια περιτροπή διαδικασία για να προσπαθήσουν να συμπεριλάβουν τα όσα κάνουν και να έχουν μια πιο συνεκτική πολιτική ε, ως αποτέλεσμα. Το δεύτερο βασικό προ, ε, θέμα είναι φυσικά η συνθήκη της Λισαβόνας. η οποία έχει πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο για την ε, ε, πολιτική για τους νέους. Δεν έχουμε επισήμως αρμοδιότητα για θέματα νεολαίας, αλλά επισήμως πλέον ε, συντονίζουμε και υποστηρίζουμε δράσεις από τα κράτη-μέλη. Η δεύτερη διάσταση, η οποία αναφέρεται στον τομέα αυτό και αναφέρεται στη συνθήκη της Δεσσαβόνας, είναι το όλο θέμα της ε, συμμετοχής των πολιτών η ε, συνθήκη δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να έχουμε συμμετοχή των πολιτών από ε, πολίτες στη δημοκρατική κοινωνία και υπάρχει δική μνήμα στους νέους ανθρώπους. Ο βαθμός συμμετοχής και ενδιαφέροντος ε, των νέων για την δημόσια ζωή είναι κάτι το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη λοιπόν το αναγνωρίζει αυτό και θα πρέπει να δούμε τι μέτρα ε, προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ε, βάσης που έχουμε από τη Νέα Συνθήκη. Και τρίτον, φυσικά, η Συνθήκη συμπεριλαμβάνει τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Για τους νέους ανθρώπους και τα παιδιά υπάρχει συγκεκριμένη αναγνώριση και προστασία και υπάρχουν φυσικά και στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τον αθλητισμό και άλλους τομείς που ενδιαφέρουν τους νέους. Το τρίτο και τελευταίο σημείο της διαφάνειας αυτής αναφέρεται στο ε, ρόλο και στις δυνατότητες που προσφέρονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η μελέτη αυτή ε, ξεκίνησε νομίζω στις αρχές της νέας δικής σας ε, προκειμένου να έχουμε και νέους προσανατολισμούς για την πολιτική για την νεολαία στα επόμενα πέντε χρόνια και με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Αβώνας και της νέας απόφασης του Συμβουλίου, οι συζητήσεις που θα κάνετε, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι καθόλου επίκαιρες. Να δούμε λίγο του τομεί δραστηριοτήτων οι οποίοι ε, μπίπτουν σε όλη αυτή τη ε, μεγάλη επικεφαλίδα της πολιτικής για την νεολαία. Ο βασικός στόχος είναι να έχουμε μία ε, πολυτομιακή προσέγγιση. Οι ανησυχίε των νέων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε πολλούς τομείς πολιτικής και εδώ η διαφάνεια ε, καταδεικνύει οκτώ τομείς ε, κοινοτικής πολιτικής στους οποίους η προσέγγιση αυτή ακολουθείται και θα επεκταθεί και περαιτέρω. Το σκεπτικό βέβαια εδώ είναι ότι όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική για την νεολαία, η Γενική Διεύθυνση δηλαδή Εκπαίδευση και Πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να συνεργαστούν με τι υπόλοιπε Γενικέ Διευθύνσει και μέσω αυτή τη διαδικασία με τι εθνικέ κυβερνήσει, τα κράτη-μέλη και τι αρμόδιε αρχέ να διασφαλίσουν ότι ε, τα συμφέροντα των νέων λαμβάνονται υπόψη στην εκπόνηση αυτών των πολιτικών. Και εδώ έχουμε λοιπόν και το mainstreaming, το οποίο χρησιμοποιείται ως κοινή προσέγγιση σε, πολλά, σε πολλούς άλλους τομείς, όπως σε θέματα ισότητας των φύλων. Εδώ θα θέλαμε να συστήσουμε Πρώτον, ότι είναι υψή τη σημασία να υπάρχουν σαφεί προτεραιότητε. Υπάρχουν οκτώ τομεί δράση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, καταρχά, να επιτύχουμε ε, πραγματική επιρροή σε όλα αυτά εάν η θέση σας είναι ότι θέλετε να ενισχύσετε απλώς ε, τα συμφέροντα των νέων, επομένως θα πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας σε κάποιου συγκεκριμένου τομείς, κυρίως να διασφαλίσουμε πολιτική δέσμευση όμως από όσου ε, έχουν τα ενία των συγκεκριμένων πολιτικών. Αν μιλάμε, για παράδειγμα, για θέματα απασχόλησης των νέων, ε, όλοι όσοι ασχολούνται με θέματα νεολαία θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με του συναδέλφου στη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τα Υπουργεία Εργασία σε εθνικό επίπεδο, για να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν πραγματικά πολιτικέ δεσμεύσει από όλου όσου ασχολούνται με αυτέ τι πολιτικέ. Και φυσικά οι ανησυχίε των νέων ανθρώπων δεν σταματούν μόνο με αυτού τους οκτώ τομεί. Επομένως ε, υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουμε και τις συνέπειες για τους νέου ε, για τις ε, πολιτικές εν γέννη πέραν των οκτώ αυτών τομέων. Τώρα, να εστιάσουμε λίγο περισσότερο. Η ανοιχτή μέθοδο συντονισμού είναι ο τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται τα κράτη-μέλη μέσω των υπηρεσιών που είναι αρμόδιε για νέου ανθρώπου και πολιτική νεολαία. Δεδομένη αρμοδιότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό, είναι κατάλληλο τρόπο εργασία. Δίνεται δυνατότητα για διαβουλεύσει μεταξύ κρατών μελών, ανταλλαγή εμπειριών, ε, δημιουργούνται κοινοί στόχοι όπου υπάρχει τέτοια δυνατότητα και διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα είναι λίγο ε, διάσπαρτα ως προς το πώς δεσμεύονται τα κράτη-μέλη και ποιες είναι οι κοινέ δεσμεύσεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, προτείνουμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα πόρων διαθέσιμων σε κάθε, σε κάθε κράτος να εστιάσουμε σε περιορισμένο αριθμό στόχων, να είναι συγκεκριμένοι αυτοί και μέσω μιας διαδικασίας όπου μαθαίνουμε ένας από τον άλλον, που είναι και η βασική προσέγγιση του Συμβουλίου, μέσω λοιπόν του peer learning, να ανταλλάξουμε καλά παραδείγματα από τα κράτη-μέλη και να τα μεταλαμπαδεύσουμε σε όλους όσους δεν έχουν την εμπειρία και τον τρόπο ίσως να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά. Αν ε, εστιάζουμε για παράδειγμα σε θέματα φύλου, προσπαθούμε να επιτύχουμε συγκεκριμένου στόχου, έτσι και εδώ θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι δείκτε που θα σα επιτρέπουν να διαπιστώσετε κατά πόσον επιτεύχθηκαν ή όχι αυτοί οι στόχοι. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν της ε, ε, διαδικασίας ανάπτυξης που έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια με την ανοιχτή ε, μέθοδο συντονισμού. Δεν έχουμε ε, ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης απόδοσης και νομίζω ότι πλέον ήγηκε και η ώρα να έχουμε αυτούς τους δείκτες ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να δουν τι πρόοδο έχουν επιτύχει μέσω της διαδικασίας. Part ε, Τέλος. Έχουμε δεδομημένο διάλογο σε αυτή την ανταλλαγή μεταξύ κρατών μελών. Όπως σας είπα και πριν, θα πρέπει να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι ίδιοι οι νέοι για την ε, δημιουργία πολιτικής και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Ο τρόπος που γίνεται αυτό και πάλι ε, ποικίλει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Ε, κάποια κράτη-μέλη έχουν μακρά παράδοση θεσμικού διαλόγου μεταξύ ε, οργανώσεων νεολαίας, εθνικών συμβουλίων νεολαίας και υπάρχουν ευθύνε και από πλευρά κυβέρνηση για πολιτικέ νεολαία και κάποιε άλλε χώρε μέλη έχουν μια πολύ λιγότερο αναπτυγμένη διαδικασία. Απόρρια του δομημένου διαλόγου είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει τη δέσμευση να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία και εδώ κάνουμε συγκεκριμένε συστάσει στον τομέα αυτό. Και πάλι υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί από πλευρά πόρων, όχι μόνο από πλευρά κυβερνήσεων, αλλά κυρίω από τι οργανώσει νεολαία. Και επομένω ε, θα πρέπει να επιλέξουμε τομεί προτεραιότητα για να υπάρχει κάποιο νόημα σε όλο αυτό και να υπάρχει μια ουσιαστική διαδικασία διαβούλευση όπου θα μπορούν να ε, συζητηθούν απευθεία τα συμφέροντα των νέων. Επίσης υπάρχει η αρχή οι μειονεκτούντε, αυτοί που έχουν λιγότερες δυνατότητες να εκφράσουν την άποψή τους και τις ανάγκες τους, να χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή. Και αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο αποτελεί μεγάλη πρόκληση για όσους κάνουν πολιτική και να επισημάνω εδώ ότι έχει επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος τα τελευταία χρόνια και φυσικά υπάρχει κάθε λόγος να το προχωρήσουμε αυτό περαιτέρω και να ε, δούμε τι πρόοδος έχει επιτευχθεί σε κάποια κράτη-μέλη και να το επεκτείνουμε όλο αυτό. Για να υπάρχει νόημα θα πρέπει να υπάρχει διάλογος όχι μόνο με αυτούς οι οποίοι ε, είναι στις πρωτεύουσε και έχουν ε, αντιπροσωπευτικό ρόλο αλλά να αναπτυχθεί και η τοπική διάσταση, να έχουμε συμμετοχή από κάτω προς τα πάνω των νέων στις οργανώσεις νεολαίας και φυσικά εδώ αναγνωρίζουμε και την αξία του να συμπεριλάβουμε με τον τρόπο τους και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει επίσημη συμπερίληψη των κοινοβουλίων σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά τα νομοθετικά και κοινοβουλευτικά όπλα στη διαδικασία θα μπορούσαν να έχουν ένα παράλληλο, παράλληλο διάλογο με τους νέους. Όλα αυτά υποστηρίζονται από πολύ μεγάλο ε, αριθμό έρευνας. Υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι ε, γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά τους νέους αν δεν ξέρουμε τις κοινωνικο-οικονομικές καταστάσεις. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένες εκθέσεις ε, οι οποίες συνόδευαν και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρχές του χρόνου και εδώ έχουμε και μια επικαιροποιημένη ε, επισκόπηση της κατάστασης της νεολαίας στα κράτη-μέλη. Η έκθεση αυτή ε, δημιουργείται από έρευνα η οποία είναι συνεχώς εν εξελίξη σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι μια πολύ σημαντική διάσταση για όλα αυτά, αλλά θα πρέπει εδώ ότι ε, η κατάσταση της έρευνας για τη νεολαία είναι άνηση Ω προ το επίπεδο και την ποιότητα των δεδομένων που έχουμε από όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό που λέμε στον τομέα αυτό είναι ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη δημοσίευση και την ε, διάδοση αυτών των πληροφοριών ε, πιο επισταμένα. Θα πρέπει να καθορίζουμε και τι δεδομένα θα πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς και αυτό αφορά και στον κόσμο της παιδείας ε, Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούνται οι εξελίξει για την παιδεία και πλέον έχει αναπτυχθεί ένα συγκεκριμένο σύστημα με βασικού δείκτε και βασικά δεδομένα τα οποία θα πρέπει να παρακολουθούνται. Ένα αντίστοιχο θα μπορούσαμε να έχουμε και για την νεολαία και έτσι η διάσταση των κρατών μελών θα πρέπει να καθορίζεται και να έχουμε έναν εναρμονισμένο τρόπο και για να ενισχύσουμε αυτή τη διαδικασία σε επίπεδο κρατών μελών θεωρούμε ότι θα πρέπει να υποστηρίξει περισσότερο η κοινότητα. Θυμηθείτε τα 900, ε, ε, εκατομμύρια των Youth ε, in Action, τα οποία έτσι καλώς θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τέλος. Ένα σημαντικό θέμα αφορά την Λισαβόνα, το ανέφερα και προηγουμένως, γιατί ακριβώς ενέχει αυτήν την έννοια της συμμετοχής και αναφέρεται τους νέους σαν μια ιδιαίτερη πρόκληση. Νομίζω πάντως ότι η πολιτικοί και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις για την πολιτική ψάχνουν ακόμα τη μαγική φόρμουλα. Δεν υπάρχει όμως τέτοια μαγική φόρμουλα υπάρχει η ενδυνάμωση αυτή της ε, ε, συνθήκης η οποία δίνει στους πολιτικούς ε, την δυνατότητα να αναπτύξουν περαιτέρω αυτό το ζωτικό, αυτή τη ζωτική έννοια. Όσον αφορά τώρα την νομική ισχύ της χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων των παιδιών κτλ. Γίνεται εδώ ε, ένα προφάιλινγκ των ε, νέων ε, και κυρίως των δικαιωμάτων των νέων στο, στο χώρο εργασίας τους. Τελευταίο σημείο να πω ότι πάρα πολλοί νέοι θέλουν να εμπλακούν στην εθελοντική εργασία και αυτό δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κάθε δικαίωμα να βοηθήσει αυτού του είδους ε, της ε, διεργασίας. Τέλος, η αναφορά της αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον αθλητισμό ε, στην ε, συνθήκη δίνει επίσης μια νέα ανάπτυξη και όθηση στον αθλητισμό. Είχα πει και στην αρχή της παρουσίασής μου ότι αυτό είναι πλέον η συνθήκη τίθεται σε ισχύ και όλα αυτά λοιπόν θα αρχίσουν να ισχύουν. Εν συμπεράσματι μπορώ να πω τα εξή, ότι τα επόμενα εννέα χρόνια είναι εννέα χρόνια πολλή δουλειά. Θα πρέπει η, βεβαίως η πολιτική να πάρουν αποφάσεις, αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί δηλαδή να, γίνει, ε, να περάσει ένα ψήφισμα από κάποιο συμβούλιο ή από κάποιους πολιτικούς. Θα πρέπει οπωσδήποτε να, δοθούν, να δοθεί συνέχεια, να υλοποιηθούν τα προγράμματα, να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια. Επίσης να πιεστούν τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να ισχύσει ο λόγος τους και να γίνει πράξη επίσης ε, να ε, ε, συμμετέχουν όλοι και στις διαδικασίες και των τριών πυλώνων. Και τέλος, όλο αυτό το μεγάλο θέμα της επικοινωνίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να, ερχόμαστε σε επαφή να, με τους νέους και σε τοπικό και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε τον κύριο Σμιτ που ζήτησε το λόγο και μετά ο κύριος Φίσερς. Ε, Ευχαριστώ πολύ για την εκτενή αυτή ενημέρωση. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση κανονικά να κάνουν μια ευρύτατη στρατηγική εθνική. Στην Ουγγαρία ε, χαράξαμε τέτοια στρατηγική και μάλιστα μέχρι το έτος 2018. Ε, από το νομοσχέδιο το Ουγγρικό. Εγώ όμως είχα την αίσθηση ότι οι πολιτικοί φτιάξανε αυτά τα σχέδια και όχι οι οικογένειες, οι γονείς, οι παππούδες ε, των ε, παιδιών αυτών. Οι πολιτικοί τι συμφέρον έχουν ε, να πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίζει και να συμμετέχει και η νεολαία στις εκλογές. Πολύ ωραία αυτά που μας είπατε, ανεξαρτησία και η συμμετοχή και τα λοιπά. Πολύ ωραία και σημαντικά, αλλά επαναλαμβάνω, αυτά όλα τα έχουν εφεύρει πολιτικοί. Εγώ θέλω μια στρατηγική που να δείχνει ότι οι νέοι ζουν κρίση αυτό τον καιρό. Δεν είδα πουθενά τη λέξη οικογένεια. Πουθενά να γράφεται. Μα οι νέοι δεν θα χτίσουν οικογένεια, δεν θα φτιάξουν οικογένεια, δεν θα αναλάβουν ευθύνη για την αηφόρο ανάπτυξη της κοινωνίας ολόκληρης. Πού είναι όλα αυτά. Θα ήθελα να δω λοιπόν ένα οικογενειακό πρόγραμμα. Η σημαντικότερη μονάδα της κοινωνίας είναι η οικογένεια. Και εκεί υπάρχει κρίση. Εγώ έχω παιδιά ε, ηλικία 40 ετών, 30 ετών και έχω και ένα εγγονάκι 5 ετών και ένα 10 ετών. Εν πάση περιπτώσει καλύπτω όλη την γάμα των ηλικιών ε, και ξέρω τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρά τα ελλείμματα που έχουμε και στις ηθικές αξίες και στην πίστη και την τονίζω την πίστη αυτή. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Θα πρέπει να ε, υπάρχει αρμονική συνύπαρξη και του μυαλού και ε, του σώματος. Πού είναι όλα αυτά στα έγγραφα. Πού είναι η ηθική διάσταση. Πού είναι η ηθική διαπαιδαγώγηση, η διάπλαση των νέων. Γι' αυτό λοιπόν πολύ συχνά οι νέοι ασχολούνται με χίλια διαφορετικά πράγματα, αλλά είναι και δική μας ευθύνη κάπου να τους ε, καθοδηγήσουμε, να τους εμφυσίσουμε την πίστη και να τους πάμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, να έχουν αλληλεγγύη, να αναλαμβάνουν ευθύνη για άλλους ανθρώπους, ε, να εργάζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάρα πολύ σημαντικό. Ούτε αυτό το βρήκα, ε, την προστασία του περιβάλλοντος, στα έγγραφα. Μια φορά λέει development, εντάξει, και for ανάπτυξη νομίζω. Αλλά θα ήθελα περισσότερο λοιπόν να έχουμε αλληλεγγύη, οικογένεια και ηθική προς αυτή την κατεύθυνση και είναι πάρα πολύ σημαντικά βέβαια αυτά που λένε τα κείμενα, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι τρεις προεδρίες τονίζουν στο πρόγραμμά τους το στοιχείο της ε, ε, συμπεριλήψης και της συμμετοχής στην κοινωνία με ε, μέσα από το πρίσμα της απασχόλησης. Εντάξει, όλα αυτά είναι καλά και σημαντικά, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι κοσμοθεωρία ε, έχουν οι νέοι, ποια είναι η ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων, τι πρεσβεύουν, τι λένε για την οικογένεια. Όλα αυτά να μας απασχολήσουν, γιατί επαναλαμβάνω η πιο σημαντική μονάδα της κοινωνίας. Εκεί νομίζω χωλαίνει πάρα πολύ το κείμενο. Nein, du hast nicht zu gesprochen, aber... Δεν εντάξει, αλλά νομίζω ότι ζητάμε πάρα πολλά από κάποιον που κάνει μια μελέτη. Ο άνθρωπος μιλάει για τα θεσμικά όργανα και τι μπορούν να κάνουν τα θεσμικά όργανα. Το περιεχόμενο να το δίνουμε εμείς. Δεν φταίει ο άνθρωπος για το περιεχόμενο. Θέλω λίγο να τον προστατεύσω και να απευθυνθώ σε εμά και να δούμε ποια είναι τα περιεχόμενα. Ο κύριος Φίσε, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι είναι πολύ δύσκολο για μια επιχείρηση τόσο δύσκολη για να βρούμε μία λύση για αυτό το πρόβλημα το οποίο είναι τεράστιο. Θα πρέπει να κατανοήσουμε τι αρμοδιότητες και τι υποχρεώσεις έχουμε εμείς ως Ευρώπη για τα θέματα αυτά τόσο ε, σε θέματα νεολαία όσο σε θέματα και σε θέματα αθλητισμού σε σχέση και με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Διότι ε, για κάποιε χώρε όπω τη δική μου τα θέματα αυτά δεν είναι μόνο κρατικέ αρμοδιότητε, είναι και θέματα των ε, αυτόνομων περιοχών. Και φαντάζομαι ότι και στη Γερμανία υπάρχει μια αντίστοιχη κατάσταση. Επομένω είναι πάρα πολύ σημαντικό να καθορίσουμε ποιο ε, κάνει τι και να καθορίσουμε και κάποιου στόχου πιο συγκεκριμένου. Θα ήθελα να προτείνω ένα στόχο Νομίζω ότι η πρόεδρος μας πρότεινε και μια επιτροπή να παρακολουθεί το θέμα αυτό, γιατί είναι η ψυχή της Ευρώπης. Να ξέρουμε ότι όλοι οι νέοι Ευρωπαίοι θα μπορούν να νιώθουν κάθε φορά όλο και περισσότερο Ευρωπαίοι, να δουν τι κοινά στοιχεία διαθέτουν οι Ευρωπαίοι, τονίζω, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, να το δημιουργήσουμε, να δημιουργήσουμε λίγο αυτή την ιδέα, αυτή την εικόνα της Ευρώπης, τα κοινά σημεία που θα μπορούσαμε να έχουμε ως Ευρωπαίοι. Και τέλος, να επιμείνω και στο θέμα συγκεκριμένων στόχων, κυρίως σε θέματα απασχόλησης ε, αυτή τη στιγμή, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερω τους νέους και ε, είναι θέμα επιβίωσης πλέον, διότι... Ε, Υπάρχει και το στεγαστικό. Υπάρχουν και νέοι που πλέον δεν μπορούν να ζήσουν ε, αλλού και ζουν πάντα με τους γονείς τους. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανεξαρτητοποίησης και να δούμε και κάποια συγκεκριμένα θέματα σε θέματα αθλητισμού. Τι μπορούμε να κάνουμε, δεν, ξέρω, δεν ήταν αντικείμενο της μελέτης, αλλά ίσως θα μπορούσε να το δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να το ανοιχνεύσουμε λίγο το θέμα, να δούμε τι αρμοδιότητες διαθέτουμε και να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, να μην μείνουμε μόνο στα ωραία λόγια. <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Ναι τη δεχτήκαμε αυτή τη μελέτη, την ακούσαμε για το περιεχόμενο και τη φορολογία, να τα συζητήσουμε. Τώρα θα ήθελα να δώσω, να δω το σημείο 8, λέει η πρόεδρο μαζί, που λέει μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΕΟΛΕ, επένδυση και δυνάμιση και κύριος Παπα-Νικολάου είναι εισηγητής μας. Έτσι και αλλιώ έχει το λόγο. Του δίνω το λόγο και για τα δύο όμω τώρα, έτσι. Και για τη δική σα πρόταση για την έκθεσή σα και για τα όσα έχετε να πείτε. Και μετά έχω άλλους δύο συναδέλφους. Παρακαλώ. Συμφωνείτε να πάρουμε και τα δύο θέματα τώρα μαζί. Παρακαλώ. Κύριε Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ. Στην... Γι' αυτό και σας ζήτησα το λόγο. Νομίζω ότι ο καταλληλότερος να προστατέψω τον κύριο Ντόχερτ είμαι εγώ για να εξηγήσω με την έρευνα που έχουμε κάνει το προηγούμενο διάστημα και προσπαθώντας να κάνω όσο καλύτερα το καθήκον μου ως εισηγητής και σε συνεργασία και με τους συναδέλφους και με πολλούς φορείς, να δούμε πέραν των τεχνοκρατικών ζητημάτων πώς μπορούμε σε πολιτικό επίπεδο το Κοινοβούλιο να συνδράμει τους νέους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Και από αυτή την άποψη θα ήθελα πραγματικά να παρακαλέσω να ε, συζητήσουμε και στο πολιτικό επίπεδο και βεβαίως μετά και ο κύριος Ντόχερτη να ε, απαντήσει στα ερωτήματα που τίθενται. Ε, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Ντόχερτη και νομίζω ότι συνέβαλε καθοριστικά στο να μην με ε, επιπλήξει στο τέλος η κυρία Πρόεδρος γιατί θα καθυστερούσα πολλά από όσα είπε ήθελα να τα πω και εγώ και θέλω να ευχαριστήσω όλο αυτό το διάστημα για τη συνεργασία που είχαμε και την Επιτροπή και το Συμβούλιο ε, το προηγούμενο διάστημα έχω συναντηθεί με του Ευρωπαϊκού Φορεί Νεολαία. Έχω ανταλλάξει απόψει με συναδέλφου. Φυσικά είχαμε συνάντηση με του κοιόδη συζητητέ, του οποίου ευχαριστώ για τη μέχρι τώρα συνεργασία. Και στα όσα υπόθηκαν, θα ήθελα ε, σύντομα να συνεισφέρω κι εγώ τα εξή. Εδώ και αρκετά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη συνθήκη του Μάστριχ και μετά έχει, ε, έχει, έχει ξεχωρίσει τα θέματα της νεολαίας και έχει δημιουργήσει διαφορετική ενότητα. Είχαμε μετά τη Λευκή Βίβλο, τα ανέφερα αυτά ο κύριος Σουντόχερτη, είχαμε το Σύμφωνο για την Νεολαία το 2005 και σήμερα ερχόμαστε με μια νέα πρόταση της Επιτροπής. Επανήλθε και το Συμβούλιο την περασμένη Παρασκευή ε, συνεπικουρώντας την Επιτροπή, καλωσορίζοντας το κείμενο της Επιτροπής και προσθέτοντας και ε, αν θέλετε μεταβάλλοντας κατά κάποιο τρόπο κάποιες θεματικές ενότητες. Η ουσία όμω παραμένει η ίδια το γεγονός ότι έχουμε αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες των οργάνων της Ένωσης και η προσπάθεια στο να εντείνουμε την έμφαση που δίνουμε στα θέματα αυτά δείχνει προφανώς αυτό που είπε προηγουμένως και ο κύριος Σμιτ και, ο κύριος Σμίτ, και αυτό που όλοι συναισθανόμαστε ότι αυτά που πρέπει να κάνουμε για την νεολαία δεν είναι αυτά που θέλουμε και σίγουρα μένουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Η ανακοίνωση ξεκινάει με τη διαπίστωση ότι η Ευρώπη γυράσκει και ο πληθυσμό τη Ευρώπη μειώνεται. <laughs> Και γι' αυτό ακριβώ όταν στο Κοινοβούλιο θέλουμε να κοιτάμε το μέλλον και θέλουμε να αναφερόμαστε σε μια καλύτερη Ευρώπη, πάνω απ' όλα πρέπει να δίνουμε έμφαση στου νέου ανθρώπου. Γι' αυτό η συζήτηση αυτή είναι εξαιρετικά επίκαιρη και πολύ χρήσιμη και το ε, διακύβευμα αυτή πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον. Αναφέρθηκε ο κύριος Ντόχερτη στις ε, θεματικές ενότητες της ανακοίνωσης Επιτροπής. Μέσα από τη συζήτηση που έχω κάνει και εγώ το προηγούμενο διάστημα και από την όσο πιο βαθιά μελέτη του θέματος, και εγώ ήθελα να αναφέρω πολλά ακόμα. Θέλαμε, για παράδειγμα, συζητώντα και με του κοιόδη συγκητέ, να δούμε πώ πρέπει να έχουμε μια ξεχωριστή θεματική ενότητα για το περιβάλλον. Έχουμε μπροστά μα την Κοπενχάγη, έχουμε πολύ σημαντικά θέματα. Ε, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να όσο μπορούμε να οριοθετήσουμε στόχους και να μπορέσουμε συγκεκριμένα και στοχευμένα κάθε φορά να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να έχουμε αποτελέσματα. Το θυμίζω ότι βρισκόμαστε ακόμη στην περιοχή της επικουρικότητας. Η συνθήκη της Λισαβόνα δίνει μεγαλύτερη έμφαση, αλλά νομικά οι αρμοδιότητες παραμένουν οι ίδιες. Για το λόγο αυτό, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι όσο μπορούμε να ενδυναμώνουμε τη φωνή μας και με τις ιδέες και τις προτάσεις και, τις, και τη συνεργασία να, μπορεί, να μπορούμε να δίνουμε υλικό στα κράτη-μέλη προκειμένου να το ενσωματώνουν. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ότι ό,τι και να κάνουμε, αν δεν υπάρχει ενσωμάτωση από τα κράτη-μέλη και δεν ε, υπάρχει έμφαση στα θέματα αυτά, δεν καταλήγουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αναφέρει η Επιτροπή, ε, επιγραμματικά λέω, τους, τις θεματικές ενότητες και μετά από κάθε θεματική ενότητα δίνει και κάποιες προτάσεις για δράσεις που πρέπει να ληφθούν. Για την, για την εκπαίδευση δεν το συζητάμε. Είναι το απαραίτητο εφόδιο για τους νέους στο μέλλον. Συζητάμε ότι οι νέοι χωρίς δεξιότητες στο μέλλον θα έχουν τεράστιο πρόβλημα. Μέσα στην οικονομική κρίση δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για την απασχόληση. Είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Να σας πω, θα, φτάσω μετά και στην έκθεση της Επιτροπής για το 2009 σε σχέση με μεγέθη και στατιστικές που υπάρχουν. Αναφέρεται στη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα, υγεία και αθλητισμός, συμμετοχή, κοινωνική ένταξη, ο εθελοντισμός, έχουμε την συζήτηση όλο αυτό το διάστημα το 2011 και του εθελοντισμού και βεβαίως οι νέοι και ο κόσμος, εννοώντα εδώ, σε αυτό το γενικό τίτλο και τα ζητήματα περιβάλλοντος και πολλά άλλα, με την έννοια ότι το περιβάλλον είναι ένα ζήτημα ε, και γι' αυτό το εντάσσουν εδώ, το οποίο αναφέρεται σε όλο τον κόσμο και δεν μπορεί σε επίπεδο κράτους μέλους μόνο να υπάρχουν συγκεκριμένες στοχεύσεις που θα φέρουν αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά σε όλα αυτά. Έχουμε την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Προσπάθησα να καταλάβω σε τι συνίσταται αυτό και πώς τελικά με αυτή τη μέθοδο καταλήγουμε σε κάτι χειροπιαστό. Εδώ έρχεται ο καθοριστικός ρόλος της Επιτροπής, εδώ έρχεται ο καθοριστικός ρόλος του Συμβουλίου και όλων ημών στο Κοινοβούλιο, με τον εξή στόχο. Πρώτα απ' όλα, να καταλάβουμε ότι σε κάθε κράτος μέλος υπάρχουν διαφορετικές δομές που δίνουν έμφαση και καθορίζουν πολιτικές για τον νεολαία. Πρέπει λοιπόν από κάθε κράτος μέλος να παίρνουμε την πληροφόρηση και τις πολιτικές που εφαρμόζονται και όλα αυτά αφού τα επεξεργαστούμε και σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες που υπάρχουν που είναι σημαντική η διατομεακή προσέγγιση όπως ανέφερε ο κύριος Δόχερτη να προσπαθούμε με, τις, με, τις, με, με τα συμπεράσματα αυτά να δίνουμε έτοιμο υλικό στα κράτη-μέλη προκειμένου και οι ίδιοι να αντιλαμβάνονται και να τους πείθουμε γι' αυτό ότι αν το εφαρμόσουν θα έχουμε αποτελέσματα. Διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτα άλλο πέραν από το να συζητάμε, να έχουμε πολύ ωραία χαρτιά. Εγώ έχω μαζέψει μια ολόκληρη βιβλιοθήκη από στοιχεία την περίοδο αυτή και συζητώντας και με την Επιτροπή πριν από δύο εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, εκεί καταλήξαμε και τους ευχαριστώ για αυτό το συμπέρασμα. <laughs> Μου είπαν οι άνθρωποι ότι πράγματι είναι πολύ σημαντικό στο επίπεδο οργάνων και υπηρεσιών έχουμε πολύ υλικό. Μου παρέδωσαν την έκθεση λέγα το 2009, θα σας πω μερικά πράγματα για αυτή μετά. Αλλά το θέμα δεν είναι να μου είπανε και συμφώνησα και εγώ απολύτως σε τεχνοκρατικό επίπεδο μόνο να έχουμε την προσέγγιση για τα θέματα αυτά. Πρέπει να έρθουν περισσότεροι πολιτικοί στη συζήτηση αυτή, οι οποίοι με την επαφή που έχουν με την κοινωνία θα μπορέσουν να βοηθήσουν περισσότερο στο να γίνουν αυτά πράξη. Και ακριβώς εδώ είναι καθοριστικός ο δικός μας ο ρόλος, διότι εμείς είμαστε το μόνο όργανο το οποίο εκλέγεται από το λαό. Εμείς λοιπόν είμαστε εκείνοι οι οποίοι πρέπει να επιστρέφουμε στις χώρες μας, να απευθυνόμαστε στους φορείς που πρέπει και σε όλους, στην ίδια την κοινωνία και να τους λέμε πάμε καλά. Και σε κάθε πολιτική που έχουμε σκεπτόμαστε ότι υπάρχουν και οι νέοι που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Γιατί δεν είναι μόνο να έχουμε μια καλή έρευνα και μια καλή έκθεση και μια καλή πολιτική για τους νέους. Αν σε κάθε πολιτική που υπάρχει για το περιβάλλον, για το ασφαλιστικό συζητάμε αυτή την περίοδο στη χώρα μου, για ε, τις μεταφορές, για την εκπαίδευση, για την εργασία. Αν σε όλα αυτά δεν λέμε ότι πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στους νέους ανθρώπους, από τη στιγμή που όλοι συνομολογούμε ότι το μέλλον της Ευρώπης είναι οι νέοι, τότε δεν έχουμε αποτέλεσμα παρά μόνο συνεχίζουμε να συζητάμε. Σε μερικά χρόνια θα έχουμε νέε πρωτοβουλίε, θα τα πούμε πάλι πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και βεβαίω έχουμε πολύ καλά προγράμματα. Βεβαίω τα προγράμματα αυτά εξελίσσονται. Το ερώτημα όμω είναι, και εγώ διαρωτώ με γι' αυτό γιατί διάβασα και τι μελέτε και προβληματίστηκα. Πράγματι, αυτοί που συμμετέχουν στα προγράμματα είναι πολύ ευχαριστημένοι. Οι άλλοι που δεν συμμετέχουν στα προγράμματα ξέρουν, καταλαβαίνουν τι πρέπει να γίνει. Αντιλαμβάνονται και βοηθάμε εμεί το να προβάλλουμε αυτή τη δουλειά στο ότι όσο περισσότερο συμμετέχουν ωφελούνται οι ίδιοι. Μου παρέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η, συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έκθεση για την νεολαία, γιατί και εγώ προσπαθούσα να βρω στοιχεία. Θα σας πω επιγραμματικά ότι πράγματι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα. Θα αναφέρω δύο-τρία μόνο ακριβώς για να εξηγήσω ότι αν σε κάτι πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στη συνέχεια για να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι υπάρχει πρόβλημα είναι να έχουμε συγκεκριμένους δείκτες, μετρήσιμους δείκτες για να εξηγούμε πώς πρέπει να δίνουμε τις προτεραιότητες. Λέει λοιπόν η μελέτη του 2009 ότι τα παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο ξεπερνάνε στο επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν λέω για κάθε χώρα γιατί υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερα νούμερα, ξεπερνάει το 15%. Είμα, και είμαστε στο 2009 και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Λέει σε ένα άλλο σημείο, τα παιδιά που είναι στα όρια της φτώχειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπου στο 18%. Λέει σε κάποιο άλλο σημείο ότι οι νέοι που έχουν ενδιαφέρον να ασχοληθούν και δηλώνουν, ε, δηλώνουν έτσι ένθερμα ότι θέλουν να έχουν μια σχέση με την πολιτική, είναι μόνο 6%. 6%. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένω αυτή τη στιγμή είναι πρόθυμοι να δώσουν σημασία σε αυτό που κάνουμε εδώ μέσα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο 6%. Δεν θα σα κουράσω. Ε, άλλο ένα στοιχείο ότι είναι αυτό που είπε ο κύριο Σμιτ για την οικογένεια και γι' αυτό το αναφέρω 37% το 2006 είναι τα μωρά που γεννιούνται εκτός γάμου. Τα λέω για να εξηγήσω ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία. Ε, περίπου το 80% των νέων στην Ευρώπη, τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν, τους τελευταίους 12 μήνες, το 80% δοκίμασε αλκοόλ και το 50% έχει μεθύσει. Και ένα τελευταίο, σε σχέση με το ίντερνετ. Σε σχέση με το 2004 έχουμε μεγάλη αύξηση της χρήσης του ίντερνετ και μεγαλύτερη εξοικείωση των νέων ανθρώπων. Υπάρχουν πολλά δεδομένα. Τα λέω όλα αυτά για να καταλήξω όσο πιο παραστατικά μπορώ, έτσι κάνοντας και εγώ μια εισαγωγή για τα θέματα αυτά, ότι με συγχωρείτε να κάνω και μια ακόμη προστίκη, συζητώντας με τους εισηγητές, κουβεντιάσαμε και για τα νεαρά άτομα με αναπηρία, κουβεντιάσαμε για τα θέματα των νέων μεταναστών και την κοινωνική ενσωμάτωση, κουβεντιάσαμε για την ανάγκη που υπάρχει να υπάρχει, αν θέλετε, μεγαλύτερη έμφαση στην έννοια της ευρωπαϊκής ιδέας και στην αξία της Ευρώπης όπως την πιστεύουμε από τα χρόνια του σχολείου, για να μπορεί ο νέος άνθρωπος να κάνει συνείδηση αυτά που κάνουμε και εδώ ερχόμαστε και επαναφέρουμε όλη τη συζήτηση σε σχέση με το ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή, με αυτά που κουβεντιάζαμε την περίοδο των ευρωεκλογών. Και καταλήγω προσπαθώντα έτσι να βοηθήσω και εγώ τη συζήτηση και να κάνουμε μια εισαγωγή ευρύτερη στο εξή. Αν εμεί έχουμε δυνατή φωνή, είναι βέβαιο και το και εγώ στη χώρα μου γιατί είχα επαφή πριν έρθω και έχω την τιμή να είμαι σε αυτό το κοινοβούλιο με τα θέματα της νεολαία, είναι βέβαιο τα κράτη-μέλη θα θελήσουν να υιοθετήσουν πολιτικές είναι βέβαιο ότι τα κράτη-μέλη θα πιστούν από τα νούμερα που σα ανέφερα. Δεν είναι δυνατόν ένα πολιτικό, ένα υπουργό που έρχεται εδώ να μην αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα πράγματα είναι συγκεκριμένα και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Είναι δεδομένο ότι στο προσεχέ μέλλον η έμφαση στη νέα γενιά πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή γιατί θα το βρούμε μπροστά μα. Κλείνοντα λοιπόν, αφού και πάλι ευχαριστήσω όλου όσου έχουμε συνεργαστεί μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουμε και λέγοντα σε όλου του συναδέλφου ότι το draft report θα είναι πολύ σύντομα. Ε, θα το έχετε πολύ σύντομα προκειμένου και εσείς να κάνετε επεξεργασία. Καταλήγω στο εξή. Το πρόβλημα δεν είναι να δώσουμε μασημένη τροφή και έτοιμες λύσεις στους νέους ανθρώπους. Το πρόβλημα είναι να δημιουργήσουμε τις δομές, να δημιουργήσουμε εκείνες οι συνθήκες μέσα από τις οποίες οι νέοι άνθρωποι από μόνοι τους θα έχουν τα εφόδια και θα έχουν τη δύναμη, το empower που λέει η έκθεση και είναι πολύ σωστό να προχωρήσουν στη ζωή, να πάρουν πρωτοβουλίες και να σταθούν στα πόδια τους. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη ενσωμάτωση πολιτικών και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή όλων των ε, βουλευτών, των συναδέλφων σήμερα εδώ, όλων των φορέων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, θα μπορέσουμε να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Είναι δεδομένο ότι είναι πολλά αυτά που έχουν να γίνουν. Πολλά, ε, νομίζω, θα, σημαντικά πράγματα θα υποθούν και σήμερα. Με πολύ χαρά θα τα ακούσω και βεβαίως θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη και για την έκθεση που από την πλευρά μας νομίζω πρέπει να υποβάλουμε. Και επαναλαμβάνω ότι η πιο σημαντική συνδρομή που μπορούμε όλοι μας να συνεισφέρουμε είναι με τη φωνή μας όλα αυτά τα σημαντικά δεδομένα, όλα τα σημαντικά αυτά που λέμε που θα τροποποιήσουμε και θα εξελίξουμε να τα ε, φωνάζουμε στα κράτη-μέλη για να τα εφαρμόσουμε. Αν δεν τα εφαρμόσουμε παραμένουμε σε πολύ ωραίες συζητήσεις, θα είμαστε ικανοποιημένοι ότι συζητάμε για τους νέους αλλά θα μένουμε μέχρι εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Γιώργο για τη μεγάλη σου δέσμευση και προσήλωση. Στις 25-26 νομίζω θα μας κάνεις ένα σχέδιο έκθεσης και θα το ξανασυζητήσουμε, ή Ιανουαρίου έτσι, ε, και συνεχίζουμε τώρα τη συζήτηση. Κυρία Μανέσκου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Ντόχερτη για τη μελέτη του, να συγχαρώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρωτοβουλία να εκπονήσει μια στρατηγική για τους νέους. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το γεγονός ότι αναφέρεται ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε συζητήσει ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναφερόμαστε στο δομημένο διάλογο για να έχουμε μία ε, διατομιακή πολιτική για τους νέους, ε, για τα θέματα που αφορούν στην νεολαία και κοιτάμε και τα θέματα τα οποία μας ανέφερε ο εισηγητής για να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη των νέων για τις αποφάσεις ε, και για να υπάρχει και ε, συμμετοχή στις πολιτικές αποφάσεις. Και ακριβώς αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, η συμμετοχή των νέων στην ε, προβληματική ε, για τα θέματα της νεολαίας που θα μπορούσαν να άπτονται όλων των ε, τομέων της πολιτικής. Θα ήθελα να σας πω ότι θα ήθελα αυτά τα συμπεράσματα και αυτά τα, ε, οι αποφάσεις που θα καταλήξουμε να μην μείνουν απλά μεγάλα λόγια, να κοιτάξουμε να δούμε πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε όλες αυτές τις στρατηγικές για τους νέους, λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς αυτές τις έννοιες, τον δομημένο διάλογο και ε, να ενσωματώσουμε τις πολιτικές ε, την πολιτική για την νεολαία σε όλε τι πολιτικέ. Θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία όπω είχαμε και μέχρι τούδε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε ε, στις πολιτικές που θα ετοιμάσουμε βάσει αυτή τη στρατηγική ακριβώ εκείνα τα στοιχεία τα οποία όχι μόνο είναι ενδιαφέροντα, αλλά είναι ζωτική σημασία για του νέου τη Ευρώπη. Και νομίζω ότι από αυτή την προοπτική μία προ, ε, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι τα ακριβή αποτελέσματα τα οποία είχε η οικονομική κρίση για τους νέους. Διότι ξέρουμε ότι οι νέοι ήταν από αυτούς που επηρεάστηκαν πολύ περισσότερο από την οικονομική κρίση και από εκεί και πέρα θα πρέπει να θέσουμε ως προτεραιότητα τα μέτρα με τα οποία θα μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τους νέους ε, ε, να λάβουν αποφάσεις, να συμμετέχουν στην αργορά εργασία και να τους δώσουμε τα μέσα για να μπορέσουν να συμμετάσχουν όλα οι τομεί είναι πάρα πολύ σημαντικοί, αυτό είναι σημαντικό, αλλά αυτή τη στιγμή ίσω πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε, αυτή, αυτό. Και να πω ότι, όπως είπα και πριν, ελπίζω ότι η στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα μας βοηθήσει να βρούμε ποιε είναι οι προτεραιότητες για τους νέου. ε, λαμβάνοντας υπόψη και όλες αυτές τις γενναιόδερες δηλώσεις ε, ε, που κάναμε και με τις οποίες συμφωνώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα οι συνάδελφοι που θα μιλήσουν τώρα να είναι και σύντομοι και να ε, απαντούν και στον εισηγητή. Μην μιλάτε μόνο για τη μελέτη και τον κύριο Ντόχερτη και αυτά που είπε ο κύριος ε, Γιώργος Παπα-Νικολάου προηγουμένως. Ο κύριος Τσμέρ παρακαλώ. <clears throat> Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για νέους πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είπαμε ότι η κοινωνία μας γυράσκει και επιβάλλεται να έχουμε πολιτική για την νεολαία. Η πολιτική της νεολαίας και η νεολαία γενικότερα δεν είναι κάτι που ανήκει σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Είναι διατομεακό, είναι κάτι το οποίο διαπερνά εγκάρσια ολόκληρη την πολιτική, παντού. Σήμερα οι νέοι, όπως ακούσαμε προηγουμένως, είναι εκείνοι που πλήττονται περισσότερο από την κρίση ακόμα και πριν εμφανιστεί η κρίση, οι νέοι εκπροσωπούσαν μια κοινωνική ομάδα πιο ευάλωτη από τις άλλες. Είχαμε πολλά αρνητικά φαινόμενα μεταξύ των νέων. Σε πιο έντονο βαθμό τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται στους νέους από ό,τι σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Λοιπόν, η ευρωπαϊκή πολιτική για την Ελλάδα θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Παράδειγμα, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε οι νέοι να βρουν δουλειά ή να βρίσκουν δουλειά καλύτερα. Και μιλώ κυρίως για την πρώτη θέση απασχόλησης. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε να εγκαταλείπουν ε, λιγότεροι νέοι το σχολείο. Να, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτό το θέμα της σχολικής διαρροής. Πώς μπορούμε να βοηθούμε τους νέους να εντάσσονται καλύτερα στην κοινωνία. Αλλά θα πρέπει να συνεννοηθούμε για το εξή θέμα και να καταλάβουμε ότι θεσμοί, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν μπορούν να επηρεάσουν τόσο πολύ τους νέους ε, στις διάφορες κοινωνίες. Γι' αυτό μιλάμε για την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Δηλαδή, οι ε, βασικοί φορείς εκεί δεν είναι μόνο τα διάφορα κράτη-μέλη, ε, ούτε τα Υπουργεία Νεότητας που είναι αρμόδια στις χώρες, αλλά υπάρχουν και σωματεία, ενώσεις, τοπικοί φορείς τοπική αυτοδιοίκηση ούτε βοηθάμε τους νέους ηθικολογώντας. Και οι νέοι έχουν ευθύνη στην κοινωνία. Και εμείς υπήρξαμε νέοι και είχαμε ευθύνη και υπεύθυνη στάση απέναντι στην κοινωνία. Οι νέοι αντιλαμβάνονται με άλλο τρόπο τις αξίες που διέπουν και εμάς. ίδιες αξίες έχουμε στην ουσία. Περίπου. Είναι γεγονός ότι σήμερα αυτή η κρίση αξιών εμφανίζεται σύμφωνα με ορισμένους, ε, κυρίως μεταξύ των νέων. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη θέση. Το Κοινοβούλιο σίγουρα πρέπει να συμμετέχει, γιατί σήμερα γίνεται διάλογος μεταξύ του Συμβουλίου και των νέων και οργανώσεων νέων. Θα πρέπει να συμμετέχουν και μέλη της Επιτροπής μας σε αυτές τις συναντήσεις, Επιτροπής Πολιτισμού και νέο Δελειώνω, Πρόεδρε. Είμαι πολύ ικανοποιημένο με την έκθεση αυτή του κυρίου Παπα-Νικολάου. Θα μελετήσω σε βάθος τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το επόμενο διάστημα, τα επόμενα ένα έτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Κύριε συνάδελφε. Ε, σε αντίθεση με εσά, εγώ είμαι υπέρ του υγιούς εγωισμού εμάς των ηλικιωμένων. Αν δεν φροντίσουμε εμείς για τους νέους μας, αν δεν το κάνουμε για λόγους λογικής, να το κάνουμε για λόγους εγωιστικούς. Η πολιτική τη νεολαία λοιπόν είναι σε πολύ καλά χέρια και αν δω και τι αποφασίζει το Συμβούλιο έχω την εντύπωση ότι το έχετε καταλάβει κι εσείς. Ε, λοιπόν, να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Χίρσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις προτάσεις αυτές. Το έγγραφο αυτό είναι πάρα πολύ εκτενές. Ευχαριστώ και τον εισηγητή μας, ο οποίος ήταν ε, σε επαφή από νωρί με εμά του σκιώδει συζητητές ε, Θα ήθελα να σας πω ότι είναι σημαντικό να αφιερώσουμε χρόνο στο έγγραφο αυτό στη συζήτηση. Είναι όλο και πιο λίγοι οι νέοι λόγω της γύρανσης του πληθυσμού, αλλά όπως το είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, παρόλα αυτά είναι στο συμφέρον όλων μας. Και αυτοί οι λίγοι νέοι που έχουμε να ε, έχουν την προσοχή που τους αξίζει. Διάβασα λοιπόν τα έγγραφα και την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα εξή τρία συμπεράσματα είναι για μένα σημαντικά. Και είναι σημαντικά για να δούμε και τι πρόοδο θα έχει η στρατηγική για την νεολαία για να κρατήσει. Το πρώτο είναι η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων, που είναι πολύ διαφορετική. Η πολιτική για την νεολαία δεν ασκείται μόνο στα σχολεία και στα κέντρα νεότητα, όπω λέει και εδώ στο έγγραφο, αλλά και σε θρησκευτικέ κοινότητε, σε αθλητικά σωματεία και συλλόγου. Και όλες αυτές ε, οι συμφωνίες πρέπει να είναι αντικείμενο συζήτηση και με αυτού του φορεί. Γιατί καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι κάθε φορέα βλέπει τον εαυτό του σε ανταγωνισμό με του άλλου. Όχι. Να πούμε ότι εδώ χρειάζεται κοινή προσπάθεια, συνεργασία. Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι Ακριβώς, ότι είπαμε η νεότητα είναι θέμα εγκάρσιο που διαπερνά τα πάντα. Δεν είναι μόνο θέμα της Επιτροπής Νεότητας, αλλά είναι και της Επιτροπής Υγείας και της Επιτροπής Απασχόλησης και δεν ξέρω ποια άλλη επιτροπή. Να λέμε και στους συναδέλφους να έχουν πάντα στο μυαλό τους και τους νέους. Θυμάμαι πριν από λίγες εβδομάδες στην Επιτροπή Απασχόλησης μια ψηφοφορία για τα μικροδάνεια τα λεγόμενα, τις μικροπιστώσεις. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι έτσι ανοίγεται και μια ευκαιρία για τους νέους αλλά δυστυχώς το έβγαλε αυτό το κοινοβούλιο, το διέγραψε στη πρόταση του. Και πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό, ε, να το λέμε και στους συναδέλφους, είναι ένα θέμα που διαπερνά όλες τις πολιτικές. Και ένα τρίτο που ακούστηκε και προηγουμένω είναι το θέμα των δικτών. Μπορούμε να γράψουμε όσα έγγραφα θέλετε και να βάλουμε όσου στόχου θέλετε, αλλά όλα αυτά κάποια στιγμή να αξιολογούνται. Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή η πολιτική νεότητα είναι ένα θέμα ήπιο, έτσι soft. Μαζευόμαστε και το συζητάμε και τι κάνουμε για του νέου. Όχι, να βρούμε κάποιου δείκτε να είναι μετρήσιμα αυτά τα πράγματα. Πιάνουν τόπο τα μέτρα. Τι κάνουν, ε, βοηθούν, μειώνεται η εγκλημότητα των νέων, η παραβατικότητα των νέων. Τα μέτρα αυτά ε, οδηγούν σε περισσότερη απασχόληση των νέων. Έχουμε λοιπόν πολλά κοινά στοιχεία, πολλές κοινέ πτυχές και με δείκτες που σε πολλά κράτη-μέλη ήδη συλλέγονται αυτά τα στοιχεία, αλλά να είναι με στόχο προσήλωση. Ε, ε θέλω να σταθώ λίγο στο θέμα της μόρφωσης και της εκπαίδευσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι από τα σημαντικότερα θέματα γενικά η παιδεία. Το ακούσαμε και προηγουμένως. Ας πούμε, η οικογένεια που είπε κάποιος συνάδελφος, να μπορούν νέοι να δημιουργούν η οικογένεια. Αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τη μόρφωση το μορφωτικό επίπεδο. Γιατί όταν έχω μια μόρφωση α, έχω και ένα εισόδημα β, μπορώ να σκεφτώ να κάνω και οικογένεια. Ή όταν κάποιος έχει τη δυνατότητα ας πούμε, να χρησιμοποιήσει σωστά το διαδίκτυο ή τα μέσα ενημέρωσης, αισθάνεται ότι έχει άλλα εφόδια για τη ζωή. Είναι πιο ε, οργανωμένος. Για το ή τα πνευματικά δικαιώματα, ε, τη μουσική που πολλοί νέοι κατεβάζουν από το διαδίκτυο. Λοιπόν, πολύ σημαντικό εδώ το θέμα της εκπαίδευσης και της μόρφωσης και εμείς στη Γερμανία βεβαίως έχουμε και ένα θέμα, δεν ξέρω και σε άλλες χώρες φαντάζομαι το ίδιο, που έχουμε παιδιά μεταναστών ε, και να δούμε ότι υπάρχουν και άλλες στρατηγικές που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Το μάθημα στο σχολείο να γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά ανθρώπων που διαμένουν παράνομα στις χώρες μας. Υπάρχει αυτό. Είναι πάρα πολλοί λαθρομετανάστες στην Ευρώπη και αυτοί έχουν παιδιά. τα παιδιά τους ε, είναι εδώ. Δεν θα έχουν καμία πρόσβαση σε σχολείο. Όταν μεγαλώσουν τι θα τα κάνουμε τα παιδιά αυτά. Και αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να το κοιτάξουμε. Και ένα άλλο, κάτι που μου λείπει σε αυτό, είναι ακριβώς τα παιδιά και οι νέοι με αναπηρίες αυτά τα θέματα από Νωρί θα πρέπει να εντάσσονται. Η Ιταλία, ας πούμε, το κάνει πολύ καλά. Στη Γερμανία, δυστυχώς, ε, ε, έχουμε πολύ μεγάλη επιλογή στα σχολεία από νωρίς. Δεν ξέρω αν βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Εμείς στη Γερμανία έχουμε να μάθουμε από άλλες χώρες για το, το πώς ενσωματώνουμε τα παιδιά με αναπηρία στο σύστημα και τους δίνουμε ευκαιρίες. Αυτά. Αυτό το τελευταίο ήθελα να το τονίσω ιδιαίτερα και ελπίζω πάρα πολύ η στρατηγική των νέων, για τους νέους να μην παραμείνει στα πλαίσια της δικής μας και μόνο κλειστής επιτροπής, αλλά να διαδοθεί σε όλο το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Κύριος Μπόρης. Ε, κατάσταση των νέων είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην ευρωπαϊκή πολιτική και πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερο περίπλοκο, διότι είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει ένα τομέα τη ζωή που να μην αφορά του νέου. Και γίνεται ακόμα πιο ε, μεγάλο το πρόβλημα, διότι τα, ε, οι πολιτικές επιδράσεις ε, κάθε φορά χάνονται. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή. Ε, συμφωνώ με τον καθηγητή Ντόχερτη. Είναι απαραίτητο να γίνει περαιτέρω έρευνα. Θα πρέπει η μέθοδος ανοιχτού συντονισμού να μας ε, υποδείξει ποια είναι τα βασικά στοιχεία για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσες ευκαιρίες ε, εκπαίδευσης, πρόσβαση στον πολιτισμό, αθλητισμός, πρόσβαση στην πληροφορία. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένο στο θέμα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας είναι οι πλέον αρμόδιοι για να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά, διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης ε, και εξέλιξη στα θέματα αυτά. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος Παπα-Νικολάου. Οι αρμοδιότητες και τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι νέοι στην Ευρώπη. και υποστηρίζω και την πρόταση του εισηγητή για ε, συμμετοχή των νέων. Θα θέλουμε, ε, θέλουμε να έχουμε νέους που θα είναι καλά καταρτισμένοι και ευαίσθητοι προς τα διάφορα θέματα. Επομένως, θα πρέπει να επενδύσουμε και μέσω εθνικών πολιτικών στην ε, ευρωπαϊκή και πολιτική εκπαίδευση. Εάν θέλουμε να έχουμε περισσότερες δραστηριότητες από πλευρά των νέων, θα πρέπει και εμείς να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ε, μορφωθούν καταλήλως οι νέοι. Μπορεί να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες, να συμμετέχουν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, πέραν τις οικογένειες που είναι ε, αυτή η οποία διαμορφώνει αρχικώς του νέους και του σχολείου που πρέπει να δώσει κατάλληλε γνώσεις και δεξιότητες, θα πρέπει να προσαρμοστεί όλο το σύστημα θα πρέπει να μας επιτρέπει να αναλάβουμε αυτή τη δέσμευση. Και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις αποτελούν σημείο κλειδί για την περαιτέρω μόρφωση των νέων. Επομένως, η Επιτροπή μας θα πρέπει να δεσμευτεί προκειμένου να είναι επιτυχής αυτή η πολιτική. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είχαμε υπολογίσει ότι θα ζητούσαν τόσο πολύ το λόγο από την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Έχω άλλους τρεις τώρα και θέλει να μιλήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το καταλαβαίνω και αυτό. Έχουν έρθει, έχει έρθει εκπρόσωπος του Συμβουλίου και περιμένει μισή ώρα να μας μιλήσει για το επόμενο θέμα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Την άλλη φορά πήρατε το λόγο νωρίς, τώρα θα χρειαστεί ίσως να περιμένετε λίγο παραπάνω. Ζητώ συγγνώμη κύριε Σελίν, παρακαλώ τους συναδέλφους να περιοριστούν στο ένα λεπτό αν μπορείτε. Ζητώ συγγνώμη. Η κυρία Παλιαδέλη παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, να δηλώσω καταρχήν ότι πολύ με ενοχλεί ίσως επειδή δεν είμαι πια νέα, να μιλώ για νέους αν πρόκειται για μια διαφορετική κατηγορία στην κοινωνία μας, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι είναι και λίγο εγωιστικό ε, ότι μιλούμε για τους νέους με δεδομένο ότι είναι το μέλλον της Ευρώπης και της κοινωνίας μας. Συμφωνώ με σε πάρα πολλά με όσα διατύπωσε γραπτά ο κ. Ντόχερτη στη μελέτη του και βεβαίως και με τον συνάδελφο στην Επιτροπή αυτή, ε, κύριο Παπα-Νικολάου, εισηγητή για την στρατηγική της νεολαίας. Μεταφέρω εδώ πολύ σύντομα την προσωπική μου εμπειρία ως δασκάλου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ως καθηγητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαπιστώσεις που δηλώνουν ότι οι νέοι, η Ευρώπη γυράσκει επειδή οι νέοι είναι απογοητευμένοι από τους θεσμούς μας. Και σε αυτό είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Διαπιστώσεις που, αφορούν ότι, που, που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι νέοι δυσπιστούν απέναντι στο κράτος, στην εξουσία. Και γι' αυτό είμαστε πάλι εμείς συνυπεύθυνοι. Διαπίστωση που αφορά στην άρνησή τους να συμμετάσχουν στα κοινά. Και αυτό φάνηκε πολύ καθαρά στην μεγάλη εποχή τους από τις πρόσφατες ευρωεκλογές. Μία τάση που, για την οποία πάλι φταίμε όλοι μας, ότι είναι αποπροσανατολισμένη και σε έναν βαθμό σε αυτό, αυτό οφείλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προβάλλει μοντέλα ε, πρότυπα αντιπαραγωγικά, αντικοινωνικά και μη συμμετοχικά. Η άρνησή τους για την ομαδικότητα, η πρόθεσή τους να δουλέψουν ατομικά και να προβληθούν σε ομαδικό και όχι σε συλλογικό επίπεδο. Και βεβαίως η ανεργία η οποία είναι το αντικειμενικό ε, ζήτημα στο οποίο μπορεί κανείς να φορτώσει όλα τα προηγούμενα. Εκτιμώ λοιπόν από το σύνολο της έκθεσης και από όσα υπόθηκαν προφορικά από τους συναδέλφους πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως τώρα παράσχει τη δυνατότητα για να δούμε αλλιώτικα οι νέοι αυτό το πρόβλημα, τα προβλήματα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι. Επομένως η ενίσχυση των προγραμμάτων Κομένιους, Εράσμος, Γιουροσκόλα, Γκρούντβιχ είναι πολύ σημαντική για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και βεβαίως η ε, προσθήκη του αθλητισμού και του εθελοντισμού στο πρόγραμμα της, ε, της στη συνθήκη της Λισαβόνας είναι επίσης πολύ σημαντική. Θεωρώ λοιπόν το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πείσουμε τα κράτη-μέλη και τις τοπικές κοινωνίες να δράσουν. Είναι δικό τους το πρόβλημα καταρχήν και η Ευρώπη είναι εδώ για να τους υποστηρίξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σκέλη. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, πρέπει να πω ότι έχει κάνει καλή δουλειά ο κύριος Στόχερτη. Προσπάθησε να εστιάσει σε ένα θέμα, γιατί είναι τεράστια ε, ε, τα πεδία που πρέπει να καλύψει. Ε, μίλησε για στόχους και για διαδικασίες μετρήσιμες, για να δούμε πώς αποδίδουν τα μέτρα. Και, και πραγματικά Εμεί θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι τέτοια τα μέτρα ώστε να ανταποκρίνονται στα κριτήρια. Επειδή μα ζητήσατε να είμαστε σύντομοι, μια μελέτη στη δική μου χώρα πέρυσι έδειξε ότι για τους νέους ε, κάτω των 25 ετών 45% δεν είχαν πάει ποτέ να ψηφίσουν. Κοιτάξτε τι απόσταση. Επίσης, ο αθλητισμό χαίρομαι που τον έφεραν και άλλοι ομιλητέ, ιδιαίτερα τώρα στη Λισαβόνα έχει μεγάλη σημασία. Με τον αθλητισμό μπορούμε να κάνουμε μεγάλη πρόοδο και να φτάσουμε στου ανθρώπου, στον εθελοντισμό, ζητήματα οικογένεια που είπε ο κύριο Σμιτ ε, και άλλα θέματα ηθικά και δεοντολογικά. Αλλά πρέπει να σα πω ότι όταν ψηφίσαμε στο Κοινοβούλιο για να γίνουν intergroup στι διακοινοβουλευτικέ ομάδε, στη δική μου ομάδα, ε, απογοητεύτηκα πολύ γιατί θεώρησαν άλλες, άλλα intergroups 14 πολύ πιο σημαντικά από τον αθλητισμό. Ε, κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Έρχεται ο Σάντα Κλάους, έρχεται ο Άγιος Βασίλης, ο Άγιος Νικόλαος, δίνουν ε, δώρα ε, και δώρα που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό. Ε, όχι μόνο ηλεκτρονικά και άλλα, ρακέτες, ε, μπάλες. Χαίρομαι λοιπόν που ο κύριος ε, Ντόχερτη τη μίλησε και για τον αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία για μας που δεν Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόεδρος. Το Γενάρη θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε και την έκθεση του Γιώργου του παπα Τώρα πολύ σύντομα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και θέλουμε να είμαστε και ευγενείς απέναντι στον κύριο Σελήν κύριο Σκούρια και μετά ο κύριος Μέρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, δύο εισηγητές που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να πω ότι ιδίω αυτά που είπε ο κύριο Παπα-Νικολάου ήταν ιδιαίτερα σημαντικά, διότι εμεί εδώ μιλάμε πάρα πολλέ γλώσσε, αλλά καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά όταν κάποιο μιλάει με ενθουσιασμό, με πάθο, με πραγματική διάθεση να εμβαθύνει σε κάποιο πρόβλημα. Όταν μιλάμε για νέου, μιλάμε για τα πάντα, γιατί μιλάμε για σχολεία, για πανεπιστήμια, για δουλειά, για οικογένεια. Και εγώ νομίζω ότι, για να συμφωνήσω και με τα όσα είπαν οι, οι προηγούμενοι συνάδελφοι, ε, θα πρέπει να εστιάσουμε όχι σε λιγότερα πράγματα, αλλά σε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να δώσουμε ως κατευθυντήρες γραμμές ε, στις ε, ε, χώρες μέλη μας. Εδώ μπορούμε να παίξουμε αποφασιστικό ρόλο, διότι μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν συγκεκριμένε πολιτικέ. Διαβάζοντα και αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς δεν μπορούμε παρά να λάβουμε υπόψη μα, για παράδειγμα, όλα τα θέματα που αφορούν ε, τους νέου με αναπηρία. Και μιλάω για πρόσβαση στην παιδεία και στην κατάρτιση, όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και στα πανεπιστήμια. Εάν ε, τα παιδιά με αναπηρία δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν από ακοδημαϊκή σκοπιά, δύσκολα θα μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνία στο μέλλον. Σας κάνω ένα παράδειγμα κοινότοπο μεν, <laughs> αλλά σκεφτείτε όλα τα κοφά παιδιά, τα οποία δεν έχουν ε, δυνατότητα να καταλήξουν πολύ εύκολα σε πανεπιστημιακές σπουδές. Αναφέρομαι επίσης και στη βοήθεια για τους νέους για να δημιουργήσουν οικογένειε ε, πρόσβαση σε πίστοση για νέες ε, κοπέλες, μητέρες. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε συμβουλές εντός εισαγωγικών στα κράτη μας. Τέλος, ένα από τα προβλήματα τα οποία επισημαίνεται και στο, στην ανακοίνωση αφορά τη λεγόμενη έννοια του κατάλληλου τρόπου ζωής, του υγιούς τρόπου ζωής. Ξέρετε ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αύξηση των, ε, της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, ε, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα διατροφής, κυρίως ε, για τις γυναίκες <coughs> και νομίζω ότι από αυτής της πλευράς δεν αρκεί μόνο το να κάνει κάποιος αθλητισμό, το οποίο εντάξει είναι βασικό στοιχείο, αλλά θα πρέπει να εργαστούμε και να προσέχουμε λίγο και τι λέμε, διότι όταν μιλάμε για κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών σημαίνει ότι λαμβάνουμε υπόψη μόνο την κατάχρηση. Σε κάποιες φορές θα πρέπει να καταδικάζεται ακόμα και η ίδια η απλή χρήση. Ευχαριστώ. Κύριο Μέρε, παρακαλώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόμου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να δώσω ορισμένε απαντήσει. Καταρχήν ξεκινάω με την παρατήρηση του Αντιπρόεδρου του κ. Σμιτ σχετικά με το εξή. Δεν πρέπει να είναι πολιτική που διαμορφώνεται από του πολιτικού, αλλά να βασίζεται στι ανάγκε των νέων. Πρέπει να γνωρίζετε ότι θα έλεγα ότι κάναμε το καταδύναμιν, αλλά σε πολλές χώρες συγκεντρώσαμε πάνω από 40.000 νέους. Είναι μια ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω του διαδικτύου και δόθηκαν χιλιάδες απαντήσεις. Εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Νοέμβριο του 2008, δηλαδή πέρσι, την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας οργανώσατε μια μεγάλη ακρόαση για το τι περιμένουν οι νέοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη δεκαετία προτιθέμεθα να συνεχίσουμε αυτό το περίφημο διάλογο με τους νέους. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να πούμε το να συζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλους τους νέους, να τους οργανώσει, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είναι εύκολο δεν πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχετε μπροστά σα. αυτή η νέα στρατηγική για να επενδύσουμε και να ενδυναμώσουμε, investing and empowering, χωρίς ε, είναι τα αποτελέσματα της ευρείας διαβούλευσης με τους νέους. Αυτή ήταν η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση, επί της ουσίας, επί του περιεχομένου δηλαδή, προτείνουμε οκτώ προτεραιότητες, αναφέρθηκε. Πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Η συμμετοχή των νέων είναι κάτι το απαραίτητο, είναι και μια νέα αρμοδιότητα στη συνθήκη που προβλέπεται με μια φράση που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διευκολύνει ε, τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Αυτή είναι μια καινοτομία τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Τώρα, ο θελοντισμό. Αυτό το μόνο ε, ε, θετήθηκε την περασμένη εβδομάδα ε, σχετικά με την, το Ευρωπαϊκό Έτος ε, θελοντισμού για το 2011, πολύ σημαντικό για τους νέους, δημιουργικότητα, κουλτούρα, δεν θα πω σε εσάς πόσο σημαντικός είναι ο πολιτισμός ε, και η κουλτούρα. Αναφέρθηκε πολλές φορές, οι νέοι στον κόσμο, η συμμετοχή των νέων στις κλιματικές αλλαγές, στην εξοικονόμηση ενέργειας και ούτω καθεξής, αυτά είναι πολύ σημαντικά, πρέπει να κινητοποιήσουμε τους νέους. Και κατόπιν έρχεται το πιο δύσκολο στάδιο, η απασχόληση, η κρίση που αναφέρθηκε από την κυρία Μαλέσκο. Πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά οι νέοι ε, στην ε, εκπαίδευση και οι νέοι που εγκαταλείπουν το σχολείο, που δεν πρέπει να του αφήσουμε στο έλεος τους. Υπάρχει και τόσο πολύ φτώχεια ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους στην Ευρώπη. Η υγεία αναφέρθηκε σήμερα, σήμερα είναι η 25η επέτειος της ανακάλυψης του ιού του AIDS. Όλα αυτά βλέπετε λοιπόν είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, εδώ επί της ουσίας σκεφτήκαμε πολύ για να υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις στο μέτρο του δυνατού. Έρχομαι στο συμπέρασμά μου. Τι θα επιθυμούσα και τι περιμένω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι περιμένουμε από εσά, υποστήριξη ε, για τις προτάσεις της Επιτροπής, ε, να μα... εμπλουτισμό θα έλεγα. Η διαδικασία είναι μακρά, η διαδικασία είναι μακρόπνοη, τρεις φορές τρία χρόνια, τρεις τριετίες. Βρισκόμαστε στην αρχή και οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικές. Επίσης αναφέρομαι και στην ομιλία του Προέδρου Μπαρόσου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου ανήγγειλε μια νέα πρωτοβουλία Europe, ε, Youth in the Move, η νεολαία εν κινήσει. Εμείς έχουμε στο νου την κινητικότητα. Έρασμος, οι μαθητευόμενοι, οι νέοι θελοντές, οι καλλιτέχνες, οι αθλητές. Κινητικότητα. Αλλά και κινητοποίηση των νέων και κινητοποίηση των πολιτικών για τους νέους. Είμαστε σε μια νέα εξέλιξη αυτής της δέσμευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία. Τώρα, η υλοποίηση, η εφαρμογή. Εδώ τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Εδώ ειλικρινά θα ήθελα να μας βοηθήσει το Κοινοβούλιο, επειδή η εφαρμογή, η υλοποίηση υπόθηκε από πολλούς, εξαρτάται από τα κράτη-μέλη. Και μάλιστα ο κ. Φίσασμπαρ το ανέφερε. Μερικέ φορέ εξαρτάται από το περιφερειακό επίπεδο. Επί Ισπανική Προεδρία θα οργανώσουμε μια διάσκεψη για να δούμε πώ μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική με τη βοήθεια ε, των τοπικών αρχών, των περιφερειών. Οι δείκτε όπου τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να έχουν δείκτε. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Εάν θέλουμε να έχουμε μια πραγματική πολιτική, χρειαζόμαστε και δείκτε. Θα ήθελα να σα πω ότι μπορείτε να στηρίζεστε στη βοήθεια της Επιτροπής, ε, κυρία Πρόεδρε, ο εισηγητής ο κύριο Παπα-Νικολάου και ήθελα να σας πω ότι παρόλα αυτά είμαι αισιόδοξο ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα πολλά για τους νέους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μερέσα. Όπως υπήρξατε πάντοτε, είστε αισιόδοξο, γι' αυτό φτάσαμε εκεί που έχουμε φτάσει και πιστεύω ότι αυτή είναι μια καλή στιγμή για να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας υπέρ των νέων, της νεολαίας και νομίζω ότι η Επιτροπή ε, συμφωνεί, ακολουθεί και εμείς το ίδιο. Πολύ καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Σήμερα συζητήσαμε πολύ καλά. Έχω την εντύπωση ότι η Επιτροπή είναι πραγματικά δεσμευμένη στο να κάνει καλή δουλειά. Τώρα θα δούμε πώς το Συμβούλιο Υπουργών μπορεί να μας βοηθήσει και μας και την Επιτροπή. Ο κ. Σιδίν, κ. συγχαρητήρια, επειδή νομίζω ότι μόλις γίνεται πατέρας μιας τρίτης κόρης. Την τελευταία φορά που βρισκόμασταν, που βρισκόσασταν εδώ, δεν είχε έλθει ακόμα στον κόσμο. Λοιπόν, να σας ζήσει, συγχαρητήρια στη σύζυγό σας να σας ζήσει μικρή. Και τις εύχομαι πολύ καλά νιάτα και στη Σουηδία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ να μας προσήσετε σε συντομία τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών ε, για τον πολιτισμό, Συμβουλίου Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μου θυμίζω την τελευταία φορά που ήμουν εδώ στην Επιτροπή σας ε, τι τρέχαμε στο γιατρό για να κάνουμε ένα check-up ε, για την εγκυμοσύνη. Ναι, είναι ένα κοριτσάκι, είναι το δεύτερο κοριτσάκι που έχω, τώρα έχω ένα γιο και δύο κόρες. Ε, όταν ακούω λοιπόν τους πολιτικούς ή άλλους που μιλάνε για τις μελλοντικέ γενναίες, σκέφτομαι τα δικά μου τα παιδιά, όπως και οι υπόλοιποι φαντάζομαι. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ. Θα ήθελα να σας εξηγήσω ότι θα σας μιλήσω για το Συμβούλιο της Παρασκευής, θα σας μιλήσω για το σκέλος, το πολιτιστικό και οπτικοκουστικό. Στέφθηκε με επιτυχία το Συμβούλιο, όλα όσα είχαν σχεδιαστεί εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια ε, ε, του Συμβουλίου, το σκέλος και εκπαίδευσης ε, και νεολαίας. Αλλά θα σας μιλήσω για τα τέσσερα σημαντικά σημεία της ημερής διάταξης όσον αφορά την, τον τομέα των πολιτιστικό και των οπτικοακουστικών. Είχαμε τέσσερα βασικά σημεία στην διάταξη. Δύο συμπεράσματα του Συμβουλίου για την πρόθεση μια δημιουργική νεολαία, κατόπιν ε, η γνώση σχετικά με το ΜΜΕ, μία απόφαση για ε, τις ε, εθελοντικές δραστηριότητες 2011 και μια ε, μεγάλη σημαντική πολιτική, ψηφιακή ε, εφαρμογή του πολιτισμού εστιαζόμενη στα βιβλία. Μετά, κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι υπουργοί συζήτησαν για ε, την ε, μελλοντική διακυβέρνηση και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής. Θα σας μιλήσω για τα τέσσερα σημεία της Ευρωπαϊκής Διάταξης, διότι γνωρίζω ότι ενδιαφέρουν τη δική σας την Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την πρόθεση μιας δημιουργικής ε, γενεάς. Ουσιαστικά αυτό αφορά τη δημιουργία, την πρόθεση της καινοτόμου ικανότητος και της δημιουργικότητας των νέων με πρόσβαση στην, σε πολιτιστικά αγαθά, ας πούμε, και στην έκφραση. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία της Προεδρίας. Είχαμε την εντύπωση ότι βλέποντας τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις στρατηγικές, αλλά και τα προγράμματά της, κυρίως το πολιτιστικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα ΜΜΕ, τα παιδιά και οι νέοι δεν θεωρούνται ως μια ομάδα η οποία πρέπει να τύχει της αναγκαίας προσοχής. Είναι μια, ένα σκέλος που πρέπει να ληφθεί υπόψη ναι, όταν εκπονούνται οι πολιτικές και οι ενέργειες. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως, ο βασικός λόγος είναι ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην κουλτούρα και σε διαφορετικές πολιτιστικές εκφράσεις από μικρή ηλικία. Και αυτό είναι ένα εργαλείο σημαντικό για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της ταυτότητας των νέων, της αυτοπεποίθησης. Και επίσης, και πολύ σημαντικό, ε, αυτό συμβάλλει στη δημιουργία ικανοτήτων, δεξιοτήτων που είναι καταλητική σημασία όταν μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά ε, και μπουν στην αργορά εργασία. Βεβαίω, επίσης για να διαμορφώσουμε σωστούς πολίτες της Ευρώπης. Ε, ένα άλλο συμπέρασμα είναι ότι φέτο είναι το έτο τη δημιουργικότητα τη καινοτομία. Συνεπώ, αυτή ήταν η προσπάθεια τη Προεδρία μα να προσθέσει στη συζήτηση ε, λέγοντα τι μπορεί να κάνει η κουλτούρα για να προωθήσει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε άλλου τομεί τη κοινωνία. Αυτά τα συμπεράσματα λοιπόν, τα οποία εγκρίθηκαν ομοφόνος από όλα τα κράτη-μέλη, σημαίνουν ότι για πρώτη φορά πλέον υπάρχει ε, μια νέα προοπτική για τους νέους και τα παιδιά στα πλαίσια της πολιτιστικής πολιτικής και της πολιτικής μέσων ενημέρωσης από πλευρά Συμβουλίου. Και αυτό σημαίνει ότι τα νέα παιδιά ε, θα ξέρουν ότι οι ανάγκες τους θα ληφθούν υπόψη για να προαχθεί η κουλτούρα. Τα συμπεράσματα επίση υπογράφησαν ότι γίνεται έκκληση στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθηθεί καλύτερη πρόσβαση στην κουλτούρα και στι πολιτιστικέ εκφράσει. Κυρίω στα σχολεία, στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι ε, τα πολιτιστικά ιδρύματα στην Ευρώπη και τα κράτη-μέλη θα διδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο για την προώθηση τη κουλτούρα εν γέννη. Αυτά ήταν τα συμπεράσματα για τη δημιουργικότητα. Ένα άλλο σύνολο συμπερασμάτων υιοθετήθηκε σχετικά με τις γνώσεις στα ΜΜΕ και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα θυμάστε ότι η Επιτροπή παρουσίασε ε, μία σύσταση το καλοκαίρι και εμείς θυμόμαστε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δημοσίευσε μία έκθεση στο τέλος του 2008. Και αυτό ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία που συνέβαλαν στη σκέψη της Επιτροπής. Η σύσταση της Επιτροπής είχε ως αντικείμενο, έτσι μας είπαν, να είναι μία ε, σύσταση σε συναπόφαση με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς όμως δεν συνέβη αυτό. Το οποίο σημαίνει ότι η Επιτροπή δημοσίευσε τις δικές της συστάσεις μόνη, αλλά εμείς ως Προεδρία θεωρήσαμε ότι το Συμβούλιο θα έπρεπε τουλάχιστον να αντιδράσει σε αυτή τη σύσταση. Και αυτό κάναμε ακριβώ όταν παρουσιάσαμε ε, συμπεράσματα του Συμβουλίου πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά αυτά τα συμπεράσματα είναι σύντομα, συνοπτικά, επειδή επαναβεβαιώνουν τα όσα ήδη έχει πει το Μάιο του 2008 το Συμβούλιο, αλλά ορισμένα τα βασικά στοιχεία που υπογραμμίζουν τα συμπεράσματα αυτά, που υιοθετήθηκαν την περασμένη Παρασκευή, είναι πρώτον Όλο το Συμβούλιο πιστεύει ότι χρειάζεται να υπάρχει θετική αντιμετώπιση ε, στις γνώσεις ε, στα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν κίνδυνοι δηλαδή, κυρίως στις σχέσεις που έχουν τα παιδιά με τα ΜΜΕ, αλλά υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν και πολλά ωφέλη που μπορούν να προκύψουν από την ψηφιακή επανάσταση και όλα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν ουσιαστικό σημείο του μηνύματος. Άλλη παρατηρήση που έγινε χρειάζεται ενεργό συμμετοχή του κλάδου των ΜΜΕ όσον αφορά να βελτιωθούν οι γνώσει για τα ΜΜΕ. Συγχρόνω, το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι τα μέσα ενημέρωση είναι ανεξάρτητο φορέας στην κοινωνία και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε και το ζητούμενο είναι να υποστηρίξουμε και να αναπτύξουμε τι διάφορε πρωτοβουλίε που ο κλάδο των μέσων ενημέρωση ε, αναπτύσσει στην Ευρώπη. Αλλά το Συμβούλιο Υπουργών υπήρξε απόλυτα σαφέ, λέγοντα ότι ο κλάδο αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Κάτι άλλο ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει όταν μιλάμε για πρόθεση, είτε πρόκειται για κουλτούρα, είτε πρόκειται για μέσα ενημέρωσης. Τα συμπεράσματα λοιπόν αυτά, πέραν από την εξελισσόμενη διαδικασία, για είναι ε, ε, επιπλέον στη διαδικασία για τις γνώσεις γύρω από το ΜΕ. Δύο ακόμα Η συζήτηση πολιτικής φύσης για την ψηφιακή του πολιτιστικού περιεχομένου στην Ευρώπη, κυρίως με άξονα την ψηφιοποίηση των βιβλίων, όχι αποκλειστικά αλλά ουσιαστικά, η βάση της συζήτησης, φαντάζομαι το γνωρίζετε, είναι ότι υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως περιεχόμενο online, copyright ε, στην ε, κοινωνία της γνώσης, όπως η Ευρωπαϊκή, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Αυτοί οι πρωτοβουλίες λοιπόν αποτελούν μία από τη βάση των συζητήσεων αυτών και μία άλλη βάση της συζήτησης είναι οι γνωστές εξελίξεις στις ΗΠΑ με τα Google Books. Πολλές χώρες αντέδρασαν στα βιβλία Google και τα μέσα ενημέρωσης μάλιστα και ο τομέας των εκδόσεων ε, αντέδρασε έντονα στα Google Books. Οι συζητήσεις που είχαν οι υπουργοί την Παρασκευή δεν ήταν μια υπουργή για τα Google Books και για τα ψηφιακά βιβλία γενικά, αλλά ήταν μια συζήτηση η οποία ήταν μια συζήτηση με ανοιχτού ορίζοντες. Λίγα λόγια για τα όσα είπαν τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι η ψηφιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου, όχι μόνο των βιβλίων, είναι μία από τι μεγάλε προκλήσει τη ε, πολιτική στον τομέα του πολιτισμού σήμερα. Δεν είναι η μόνη πρόκληση, υπάρχουν κι άλλε που πάντοτε ε, υπάρχουν, αλλά είναι μία από τι ουσιαστικέ προκλήσει. Και το ζητούμενο είναι πώ μπορεί η πολιτική κληρονομιά συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων να είναι ε, προσβάσιμα στους πολίτες της Ευρώπης. Υπογράμμισαν οι Υπουργοί ότι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στην ψηφιοποίηση θα πρέπει να βασίζεται ε, σε σαφή σεβασμό του copyright, τα συγγραφικά δικαιώματα, ε, τα πνευματικά δικαιώματα γενικά, αλλά και σε μια και σε έναν υγιή και σαφή ανταγωνισμό στην αγορά. Αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία που υπογραμμίστηκαν. Η Γαλλία, ο Γάλλος Υπουργό, ο κ. Μητερό, έκανε μια πρόταση σχετικά με τις συμφωνίες μεταξύ δημοσίων φορέων και ιδιωτικών φορέων στον τομέα της ψηφιοποίησης. Ο Υπουργό δεν το ανέφερε, αλλά τα πράγματα τα οποία υπενήσονταν ήταν το γεγονός ότι υπάρχουν δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ευρώπη που έχουν συνάψει συμφωνίες με ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως η Google για την ψηφιοποίηση του υλικού τους και αυτό είναι σημαντικό. Είναι ένας τρόπος για να υπάρξει μεγαλύτερη πρόσβαση. Ο Γάλλος υπουργό υπεστήριξε ότι ίσως θα πρέπει να υπάρχουν γενικές κατευθυντήριες γραμμές στην Ευρώπη, ώστε πώς μπορούν αυτές οι συμφωνίες μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να δημιουργηθούν. Πολλοί υπουργοί λοιπόν στη συζήτηση της παρασκευή, υποστήριξαν την πρόταση της Γαλλίας. Η πρόταση πιθανόν θα προωθηθεί ε, από την ε, Ισπανική Προεδρία. Και μία ιδέα που διατυπώθηκε από τον Γάλλο Υπουργό ήταν να συγκροτηθεί μια επιτροπή αξιοσέβαστων Ευρωπαίων προσωπικότητων, ολιγομελής επιτροπή, η οποία θα έχει ως εντολή να υποβάλει μια έκθεση με προτάσεις για κοινέ κατευθύνσεις γραμμές ε, όσον αφορά τις ε, συμπράξει ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Τέλος, δύο λόγια για τον εθελοντισμό. Σύμφωνα με το τελικό κείμενο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, όπως γνωρίζω, συζητήσατε και πρόσφατα υιοθετήσατε μια έκθεση σχετικά. Απλά θα ήθελα να πω ότι αυτή είναι η απόφαση η οποία έτυχε ευρεία υποστήριξη. Επίση υπήρξε σαφές σε εμά ότι η κοινωνία των πολιτών, πολίτες δηλαδή, έχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες από αυτό το έτος. Εμείς στα πρώτα στάδια της θα λήξαμε σε μια συμφωνία μεταξύ κρατών μελών στο Συμβούλιο. Οι δυσκολίες δεν ήταν πολύ δύσκολες. Συγχρόνως η Σουηδική Προεδρία κατέστησε σαφές και στα κράτη-μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα θέλαμε στο μέτρο του δυνατού να έχουμε ένα κοινό έδαφος κυρίως για το θέμα της έγκαιρης έγκρισης αυτού του φακέλου. Εγώ είχα επαφές με τον εισηγητή τον κύριο Σκούρια και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και βεβαίως την κυρία Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας που ενδεχόμενα ίσως οδήγησαν στο γεγονός και το λέω, ίσως οδήγησαν στη θετική έκβαση, δηλαδή την Παρασκευή ελήφθη απόφαση για ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθελοντισμού με 8 εκατομμύρια ευρώ προπολογισμό για το έτος που ίσως δεν είναι όσα θα ήθελαν όλοι, αλλά είναι 23% περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προταθεί από την Επιτροπή. Ο λόγος της αύξησης είναι ότι μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου θεωρήσαμε ότι ήταν λογικό να αυξηθεί ο προπολογισμό που προβλέπονταν από την απόφαση. Από την άλλη πλευρά, το Κοινοβούλιο έκανε πολύ καλή δουλειά, εξασφαλίζοντα ότι η γνωμοδότηση ήδη είχε φτάσει. Αυτές, αυτά τα επιπλέον χρήματα που προσθέθηκαν, επίσης ε, μεταφράζονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η βασική έκβαση λοιπόν ε, της οπτικοακουστικής συνεδρίασης στα πλαίσια της ε, Πολιτιστικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Και την θυμίζω αγαπητοί συνάδελφοι ότι λάβαμε τον γλυκό κείμενο. Ε, Έχετε τα πρακτικά του Συμβουλίου. Πριν από μία ώρα μπορείτε να τα διαβάσετε όλα. Τουλάχιστον οι βουλευτές τα έχουν. Δεν ξέρω οι συνεργάτες, οι βοηθοί, αν θέλετε έχουμε μερικά αντίτυπα εδώ μπροστά. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Άρχεται η συζήτηση τώρα. Θα ήθελα να πω καταρχάς εγώ ότι χαίρομαι που το Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στα θέματα της ψηφιακής εποχής, της Europeana, όπως και να το λέτε, γιατί πάντα συζητάμε και για το Google, για την Europeana, καμιά φορά κατονομάζονται, καμιά φορά όχι. Διαβάζοντας όμως οι γερμανικές εφημερίδες κατάλαβαν ότι ε, υπήρξαν και θετικές συζητήσεις την Παρασκευή για την Ευρωπαϊκή και είμαστε στο μέσο της επικαιρότητα και ακόμα και το Συμβούλιο Υπουργών το κατάλαβε και ασχολήθηκε με αυτό το θέμα στις αποφάσεις. Ευχαριστώ. Τους συναδέλφους ε, παρακαλώ τώρα να κάνουν τις ερωτήσεις τους αν έχουν στον κύριο Σελήν. Ε, Όχι από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σελήν και πάλι. Και σας παρακαλώ να έχετε μαζί σας το έγγραφο αυτό. Είναι πραγματικά στο χαρτί αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε, τι μας επιφυλάσσει το Συμβούλιο για το μέλλον. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει όχι και πού μπορούμε να ασκήσουμε πίεση. Θα ήθελα να επαναλάβω ξανά, γιατί μίλησε χθε η κυρία Τούρπελ για το θέμα της βιβλιοθήκης ψηφιακής Ευρωπαϊκή. Υπάρχει μια επιτροπή που πρότεινε ο κύριος Μιτεράν για τα λεγόμενα ορφανά έργα. Τα γνωρίζετε αυτά, τουλάχιστον η κυρία Τρούπελ το βλέπει ευνοϊκά. Ε, να δούμε ε, πώς ε, θα έχουμε την Επιτροπή Σοφών, γιατί τους χρειαζόμαστε αυτούς τους σοφούς. δεν ξέρω πού τους διαλέγουμε και πώς με βάση τη σοφία τους, αλλά ελπίζω να είναι και σοφή η απόφασή τους. Ε, μπορούμε να βρούμε και στο Google και αλλού τέτοια έργα, αλλά θα πρέπει το περιεχόμενο να είναι πραγματικά αξιοπρεπές, σωστό και αντανακλά την ευρωπαϊκή ψυχή και την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Α, τώρα ζήτησαν δύο το λόγο, το φαντάστηκα. Η Χέλγα και μετά η κυρία Παλιαδέλη. Είναι πολύ ενθαρρυντικά τα πράγματα όταν μιλάτε. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το ζήτημα της ομάδας υψηλού επίπεδου. Όταν έχουμε ε, συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να γίνεται έτσι, να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει μια σαφής προσέγγιση για το ποιες θα πρέπει να είναι οι ευρωπαϊκές προϋποθέσεις για αυτές τις ε, συμφωνίες. Αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Μέχρι τώρα για τις συμφωνίες για την Google με τις μεγάλες βιβλιοθήκες έχουμε στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συνθήκη, διότι μιλάμε για μια συμφωνία με μια ιδιωτική ε, εταιρεία και επομένως είναι μυστική. Και αυτό είναι κατά την άποψή μου το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν ξέρουμε τι μπορούν να τα με αυτά τα δεδομένα. Κάποιοι λένε, αλλά δεν είναι επίσημο, διότι δεν επιτρέπεται να τα πούνε σε όλο τον κόσμο, ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα οι ίδιοι και μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν και στο διαδίκτυο. Αλλά εδώ είναι λίγο το θολό σημείο και ίσως θα μπορούσατε να μας το ε, αναφέρετε λίγο πιο ενδελεχώς εδώ τι συμβαίνει, διότι θα είναι, πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφείς οι προποθέσει. Η κυρία Παλιαδέλη. Δικαστική σχεδόν ερώτηση. Θα μπορούσε ενδεχομένω η Επιτροπή μα να εκπροσωπηθεί στην Επιτροπή Σοφών ε, ε, μήπως ένα από τα μέλη δηλαδή της Επιτροπής Σοφών θα μπορούσε να είναι ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής Πολιτισμού και θα πρότεινα την κυρία Τρούπελ η οποία είχε ασχοληθεί και με το ζήτημα. Θα ήταν νομίζω πολύ επικοδομητικό για, την, για το έργο της Επιτροπής να έχουμε μία εκπρόσωπο και μάλιστα τη συγκεκριμένη συνάδελφο. Ευχαριστώ. Δεν είμαι βέβαιη αν είναι σοφή η κυρία Τρούπελ. Ξύπνια είναι. Ε, τώρα και σοφή, όπω το φαντάζεται ο κύριο Φεντερίκ Μιτεράν, ε, επιτροπή σοφών, τολμώ να το αμφισβητήσω. Ούτε εγώ είμαι και πολλοί από εδώ, του εδώ παρόντε. Εν πάση περιπτώσει, να το σκεφτούμε όμω. Ναι, ε, καλή πρόταση. Ευχαριστώ. Το κοιτάξουμε. Κύριε Σελήν, θέλετε να το σημειώσετε, αν έχετε την καλοσύνη. Θα προσπαθήσουμε κι εμεί κάπω να προωθήσουμε αυτή την ιδέα. Να έχει ίσω και συμμετοχή το Κοινοβούλιο με κάποιον που ασχολείται εντατικά με αυτά τα θέματα και είναι και πάρα πολύ έξυπνο, χωρί να είναι απαραίτητο και σοφό, έτσι. Δεν έχει φτάσει ακόμα στην ηλικία τη Σοφία, περίμενε. Ε, και να το σημειώσουμε αυτό. Κύριο Σκούρια. Ναι, ούτε κι εγώ είμαι ιδιαίτερο σοφό, επομένω συγχωρέστε με, αλλά ήθελα να κάνω κι εγώ μια αποτίμηση για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Νομίζω ότι η απόφαση του Συμβουλίου είναι μία απόφαση η οποία μας ικανοποιεί κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, οικονομικώς είχαμε ζητήσει περισσότερα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όπως ε, είπαμε και σε κάποιες ε, συναντήσεις μας, σπανίως αυτές τις διαδικασίες επιβεβαιώνεται ο αρχικός προϋπολογισμός, ε, ούτε καν αυξάνεται. Νομίζω λοιπόν ότι επιτύχαμε καλό αποτέλεσμα διότι το μεγαλύτερο τμήμα των χρημάτων που θα έχουμε θα χρησιμοποιηθούν για τις πρακτικές εφαρμογές επιτόπου υπέρ των οργανώσεων. Από αυτή της πλευράς λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σελίμ για όλα όσα κάναμε αυτές τις εβδομάδες. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα, αλλά έγινε πολλή δουλειά και νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερο ε, ε, ικανοποιητικό και για το Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για